Il Συνεχίζουμε την ε, συζήτηση. Η έκθεση Κάλλας προς μια νομοθετική πράξη για την ε, ψηφιακή ενιαία αγορά. Να περιμένουμε να βγει και η φωτογραφία. Και χαιρετίζουμε τον πρόεδρο Γιούνκερ. ημερήσια διάταξη προς μια νομοθετική πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά. Το λόγο έχει ο κύριος Κάλλας, εισηγητής. Η κυρία Κάλλας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν στην εκπόνηση αυτής της έκθεσης, ιδίως την συνεισηγητρία, την κυρία Γκέπχαρτ και όλους τους κοιόδης εισηγητές. Είναι μεγάλη με ικανοποίηση που η έκθεση αυτή ξεκάθαρα δηλώνει ότι χρειαζόμαστε καινοτομία και ψηφιοποίηση στην Ευρώπη και τάσεται υπέρ αυτών των κατευθύνσεων. Εάν θέλουμε οι εταιρείε να καινοτομούν, πρέπει να αποστέλουμε ένα σαφέ μήνυμα ότι στηρίζουμε την καινοτομία. Οι επιχειρήσει πολύ συχνά να ακολουθούν τη σύσταση να ε, περάσουν από παραγωγή παλιότερων προϊόντων ξεπερασμένων σε νέα πρωτότυπα προϊόντα. Θα πρέπει λοιπόν όταν κάτι δεν εξυπηρετεί το σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκε να μπορούμε να το αφήσουμε και να σκεφτούμε κάτι καινούριο, ρηξικέλευθο. Είναι πολύ σημαντικά λοιπόν όσα λέει η έκθεση αυτή για την οικονομία της περιοχής Σέγγεν αλλά και για τους φραγμούς που προβλέπουν τα κράτη-μέλη με... Ε, μια τάση να παρεμποδίζουν τους εαυτούς τους αντί να υπάρχει ένα σταθερό πλαίσιο για να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι οι μεγάλες πολυεθνικές έχουν τις, ε, τα εργαλεία και τις δυνατότητες να συμμορφωθούν με πολλά διαφορετικά σύνολα κανόνων. Όμως η οικονομία της Ευρώπης βασίζεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτές πλήττονται περισσότερο από τους φραγμούς που υπάρχουν ακόμη. Περιμένω λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει δράση προκειμένου να διατηρήσει την ακαιρεότητα της ενιαίας αγοράς. Και αυτό όχι μόνο για την ε, κοινή μας οικονομία, αλλά και για το μεγάλο κύμα καινοτομίας με τα μεγαλύτερα δεδομένα και το διαδίκτυο των πραγμάτων, όπως έχει ονομαστεί. Εάν δεν ακολουθήσει μια κατεύθυνση κυβερνοασφάλειας, τυποποίησης και ελεύθερης ροής δεδομένων η Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε θα χάσουμε ένα μεγάλο μέρος του δυναμικού μας, το οποίο είναι ζωτική σημασία για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Περιμένω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εργαστεί σκληρά, ώστε το διαδίκτυο να παραμείνει μια πλατφόρμα ελεύθερη και ανοιχτή για την κοινοτομία και τις επικοινωνίες. Βεβαίως και η ενδιάμεση οι ίδιοι αμεσολαβητέ δεν μπορεί να έχουν περιορισμένη λογοδεσία. Δεν μπορεί το διαδίκτυο να κάνει τη δουλειά των ε, αρχών επιβολή του νόμου. Πρέπει να μην υπάρχει λογοκρισία και να προστατευτεί η ελεύθερη έκφραση. Και επίση πρέπει να είναι συνειδητοποιημένοι οι χρήστε. Κάτι το οποίο το επισημαίνει επίση η έκθεση. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι οι πολίτε έχουν πλήρη γνώση και μπορούν να χειριστούν την ανταλλαγή των δεδομένων του μεταξύ των παρόχων που θα μπορούν να πρέπει εύκολα να αλλάξουν. Θα πρέπει να υπάρχει όμω και ένα βασικό επίπεδο ασφάλεια, όπως η κρυπτογράφηση και η επικαιροποίηση λογισμικού αυτές ε, τις ευθύνες, αυτές, είναι δική μας ευθύνη να κάνουμε τους πολίτες να είναι συνειδητοποιημένοι. Δεν μπορούμε να πούμε πώς να ζήσουν τη ζωή τους και τι να κάνουν οι ποιες υπηρεσίες να επιλέξουν. Γι' αυτό η ομάδα μας δεν συμφωνεί με την παράγραφο 8 και ελπίζω να στηρίξουν την τροπολογία μας 24 συνάδελφοι. Διότι ε, στο κάτω-κάτω της γραφής οι πολίτες μόνοι τους αποφασίζουν ε, την δική του ζωή και αντί να τους διευκολύνουμε ακριβώς αυτή τη ζωή ε, θα πρέπει να σκεφτούμε ε, απλούστερους τρόπους, όπως με το e-government, την ηλεκτρονική κυβέρνηση. Οι δημόσιες αρχές θα μπορούσαν να ζητούν κάποια άγραφα μόνο μία φορά λόγου χάρη. Αυτό είναι ήδη μία πρώτη κίνηση. Και πολύ σωστά το Κοινοβούλιο ζητάει να εφαρμοστεί αυτό. Είναι πάρα πολλά αυτά που θα μπορούσα να πω σε, για μια τόσο ευρία έκθεση που καλύπτει ένα τέτοιο φάσμα θεμάτων. Αλλά θα σταματήσω εδώ και σα ευχαριστώ ανυπομονώ για τη συζήτηση. Πρόεδρο, ευχαριστούμε κυρία Κάλλα. Η συνεισηγήτρια, η κυρία Γκέπχαρτ. Εύελιν, έχετε το λόγο για τέσσερα λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ την κυρία Κάλλας για την πολύ καλή συνεργασία. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το ότι ε, έλαβε τόσο μεγάλη σημασία στην ομιλία σας ε, η sharing economy, ενώ στην αρχή ούτε καν σκοπεύατε να το αναφέρατε, άρα βρισκόμαστε σε μια καλή αρχή. Στον τομέα των ανακοινώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρόκειται όμως για ζητήματα τα οποία δεν καλύπτονται καθόλου. Είναι αυτά που έχουν να κάνουν με τα εργασιακά δικαιώματα, τα κοινωνικά δικαιώματα, και άλλα αντίστοιχα που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε εάν θέλουμε να προχωρήσουμε πραγματικά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πολύ σημαντικό αυτή η ψηφιακή εσωτερική αγορά να αναπτυχθεί. Να γίνει μια πραγματική αγορά χωρίς σύνορα. Όταν ο πολίτης θα μπορεί να αγοράσει κάτι πέραν των συνόρων με τους ίδιους όρους. Γι' αυτό είναι πολύ καλό το ότι ανακοίνωσε προτάσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι δεχόμαστε διαφορετική νομοθετική μεταχείριση των διαγραμμικών και μη διαγραμμικών αγορών. Απλώς θέλουμε τα ίδια δικαιώματα για τους καταναλωτές όπως και για τις επιχειρήσεις. Αυτούς επιδιώκουμε να υποστηρίξουμε και γι' αυτό ε, θα είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματεύεται τα ζητήματα αυτά. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόμαστε ακριβώ στο ίδιο μήκο κύματο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ένα θέμα και θέλουμε ιδιαίτερα να την ευχαριστήσουμε, το θέμα του γεωγραφικού αποκλεισμού, geo-blocking. Δεν είναι παραδεκτό πολίτε τη Ευρώπη να μην μπορούν να επωφελούνται τη εσωτερική αγορά επειδή δεν βρίσκονται στη σωστή διεύθυνση ή δεν έχουν τη σωστή εθνικότητα ή γιατί η πιστοτική τους κάρτα ε, προέρχεται από ε, το λάθος κράτος. Δεν σημαίνει αυτό, δεν ισοδυναμεί αυτό με ελεύθερη διακίνηση. Εδώ θέλουμε πρόοδο και βέβαια θα συνεργαστούμε εντατικά για να προωθήσουμε κάθε δυνατή λύση. Στον τομέα του ψηφιακού περιεχομένου επίσης υπάρχει σοβαρότατος κατακαιρματισμός στην Ευρώπη απαράδεκτος κατακαιρματισμός και γι' αυτό πρέπει ιδιαίτερα να μεριμνήσουμε ότι ορισμένα επιχειρησιακά μοντέλα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή δεν θα να μην οδηγήσουν σε μονοπωλιακές καταστάσεις που θα αποβούν εις βάρος της Ευρώπης. Ο πολίτης πρέπει να έχει το δικαίωμα όταν έχει ε, μια συνδρομή κάπου, όταν είναι πελάτης κάπου, να μπορεί αυτό να το εκμεταλλεύεται σε ολόκληρη την Ευρώπη, ανέξαρτος του που βρίσκεται. Αλλιώ δεν υπάρχει ελεύθερη διακίνηση, Αλλιώ διακίνηση, αλλιώ δεν υπάρχει ελεύθερη αγορά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένας άλλο τομέα, γιατί βέβαια δεν μπορώ όλους να τους εκθέσω μέσα σε τέσσερα λεπτά. αλλά επισημαίνω έναν ο οποίο μας προβλημάτισε και είχαμε αντιπαραθέσει στις τελικέ μα συζητήσεις, το θέμα της διαχείρισης, της ηλεκτρονικής διαχείρισης. Χρειάζεται λοιπόν να απλουστευθεί αυτός ο ψηφιακός κόσμος για να προχωρήσουμε. Με πιο απλές λοιπόν λύσεις, το θέμα όμως της αρχής once only, άπαξ, ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά ταυτόχρονα γεννά ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και ασφαλώς ορισμένα κράτη και συνταγματικών περιορισμών. Σε αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για να προχωρήσουμε, ναι με την απλούστευση αλλά ταυτόχρονα και σεβόμενη την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τις συνταγματικές τάξεις των κρατών μελών. Σε αυτά ξέρω ότι ακόμα με περιμένει δουλειά. Δυστυχώ εξάτλησα το χρόνο μου. Θα, έχουμε ακόμα, θα είχαμε πολλά ακόμα να πούμε για την έκθεση αυτή. Παντώ για άλλη μια φορά ευχαριστώ θερμά όλου του συναδέλφου και σκιώδη ε, εισηγητέ, ε, το προσωπικό μα ε, για τη συνεργασία, για τη συμβολή του. Και πρέπει να σας πω ότι ήταν και πολύ ευχάριστη αυτή η συνεργασία. Ακριβώς επειδή ήταν τόσο περίπλοκο το θέμα. Ευχαριστώ. Ακούσαμε τις εισηγητρίες. Χαιρετίζω για το κοινό που παρακολουθεί αυτή την τόσο σημαντική συζήτηση και τώρα από τις πολιτικές μάλλον από τι κοινοπολιτικές επιτροπέ. Από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, ο κύριο Σόρου για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι στην Επιτροπή ΕΚΟΝ. Ε, Εξετάσαμε πολύ προσεκτικά το θέμα αυτό και επιτροφήκαμε σε δύο σημεία, ε, σκεφτόμενοι και την ε, τόσο μεγάλη οικονομική σημασία του τομέα αυτή. Με 800 ε, δις ευρώ κυκλοεργασιών ετησίως, που θα μπορούσε να δημιουργήσει 3 ε, εκατομμύρια 900.000 θέσεις εργασία στην Ευρώπη. Ε, εδώ μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι όροι πρόσβασης και συνθήκες διακυβέρνησης που είναι αποτελεσματικοί για την Ευρώπη και το συμφέρον των πολιτών. Θέλουμε η Ευρώπη να είναι κυρίως ε, ψηφιακή και αυτό που ορίσαμε και ως πολιτική γραμμή το Digital First. Και βεβαίως να υπάρχει και ψηφιακή πυρολογία. Ε, δηλαδή να υπάρχει μια ομαλή πορεία στην μετατόπιση των, των εταιριών και την παροχή υπηρεσιών σίγουρα θα πρέπει να δούμε τι ψηφιακέ υπηρεσίε και από την πλευρά τη παροχή και από την πλευρά τη κατανάλωση για να είναι αποτελεσματική η προσφορά του. Επίση, όσοι δημιουργούν ε, καινοτομία, όσοι παράγουν καινοτομία με την ίδρυση νέων επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Αυτή την οικονομική ανάπτυξη θέλουμε και θα μπορούσε να λειτουργεί αυτό και ω γνώμονα, ω φάρο για τη διεθνή αγορά. Επισημάναμε επίση τον κίνδυνο νέων μονοπωλίων που θα μπορούσαν να αναδυθούν, τα οποία εύκολα μπορούν να δημιουργηθούν και μπορούν να ανθίσουν ε, επίσης εύκολα. Ε, με κερδοσκοπικές τάσεις από τους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών, ξεπέρασα το ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Στάινρουκ και για σας ένα λεπτό εκ μέρους της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εάν ε, μπορούσαμε να περάσουμε τις θέσεις της Επιτροπής μας, θα είχαμε πολύ πιο σημαντική έμφαση δώσει στα εργασιακά και τα κοινωνικά ζητήματα, αυτά τα οποία δυστυχώς δεν υπάρχουν. Και ευχαριστώ ρητά την Εύλην Γκέπχαρτ, η οποία ιδιαίτερα με ρίμνησε για τα ζητήματα και της κοινωνικής ε, ασφάλισης για τους εργαζομένους στο ψηφιακό χώρο. Αγωνίστηκε. Ε, ξέρουμε ότι η ψηφιακή μεταστροφή δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη, αλλά πρέπει να γίνουν οι αναλύσεις σχετικές με τις επιπτώσεις της ε, στο, στα επαγγέλματα για το μέλλον, στον τρόπο εργασίας στο μέλλον, ε, τις δυνατότητες για την συνέχιση λειτουργίας των ασφαλιστικών ταμείων, το θέμα της κατάρτισης του διαβίου μάθησης, το crowd working, το shared economy, όλα αυτά τα οποία ε, μόλις διαφαίνονται τώρα, αλλά για τα οποία πρέπει να προβλέψουμε νομοθετικές ρυθμίσεις ε, που θα επιτρέψουν και στο μέλλον καλές και βιώσιμες θέσεις εργασίας και στο διαγραμμικό περιβάλλον. Ευχαριστώ. Επιτροπή των Μεταφορών και Τουρισμού, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω ε, τις συζητήτρε και όλου όσου συνέφεραν στην ε, σύνταξη της έκθεσης αυτής. Χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατάφερε να καταλήξει εκείνη θέση για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα. Οι μεταφορές είναι ένας τομέας όπου μπορούμε να υποφεληθούμε πολύ από την ψηφιακή διάσταση διότι η διαχείριση των δεδομένων θα είναι περισσότερο ασφαλής, πιο εύκολη και πιο αποτελεσματική στο μέλλον. Η χρήση δεδομένων για τις μεταφορές είναι κάτι το οποίο έχει βελτιωθεί. Είχαμε τεράστια αλλαγή όσον αφορά την ζήτηση και την προμήθεια, την προσφορά υπηρεσιών μεταφορών εξαιτία των εξελίξεων στο ψηφιακό τομέα. Όσο λοιπόν προχωρούμε προς τις ψηφιακές υπηρεσίες μεταφορών, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε κοινού κανόνες που θα επικεντρώνονται στον καταναλωτή. Η κυρία Καμερέβερτ, ένα λεπτό, Επιτροπή Πολιτισμού. Ευχαριστώ. οι πολύ σημαντικές αλλαγές που προκύπτουν από την ψηφιοποίηση είναι ορατές και στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο, αλλά όχι μόνο και το κινητό τηλέφωνο έχει μεταφέρει και το διαδίκτυο έχει μεταφέρει, έχει σπρώξει τρίτη θέση προτίμησης των νέων ε, την τηλεόραση. Υπάρχουν ε, πολύ μεγάλες δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη του διαδικτύου. Εάν θέλουμε λοιπόν τόσο ο δημόσιος και ο ιδιωτικός πάροχος τηλεόρασης να παραμείνει σημαντικός για να προβάλλει και την ε, πολυφωνία και την ελευθερία της έκφρασης πρέπει να ανοίξει τηλεόραση στο διαγραμμικό περιβάλλον. Έτσι λοιπόν η σχετική οδηγία είναι απαραίτητο να κατατεθεί και να προωθηθεί. Χρειάζεται να κοιτάξουμε αυτά τα σημεία και νομίζω ότι η ψηφιοποίηση για την ε, για τον τομέα της ε, τηλεόρασης, για το δημιουργικό αυτό κλάδο πρέπει να προχωρήσει και να εξασφαλίσει μια ε, ισότιμη μεταχείριση και για τον χρήστη και για τον διαμεσολαβητή και για τον πάροχο. Χρειάζεται πολύ περισσότερη προσήλυση για την ανάπτυξη του media competence, ιδιαίτερα σε σχέση με τους νέους, αλλά και γενικότερα για όλες τις γενιές. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τζαμπάσκι για την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και εσείς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ συνάδελφε. από την Επιτροπή ε, Νομικών Υποθέσεων και ως ο για την έκθεση αυτή. ήθελα να συγχαρώ τις εισηγητές και όλη τους τη δουλειά για τον τους και αυτό. Χάρη στις κοινές μας προσπάθειες πετύχαμε ένα πολύ καλό σημείο ισορροπίας και μια στοχευμένη πρόταση πιστεύω. πετύχαμε και τις βασικές μας προτεραιότητες, την φορητότητα την οποία θα πρέπει να προωθήσουμε, αλλά υπάρχουν και άλλα ζητήματα, όπως οι κανόνες για τα πνευματικά δικαιώματα. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν μια καλή αφετηρία και ε, καθοδήγηση. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εφαρμοστεί σωστά ο κανονισμός σε ζητήματα που μπορεί να χρειαστούν περαιτέρω μελέτη. Να μην αποφασίσουμε γρήγορα, βιαστικά και προδικάσουμε την εξέλιξή τους. Πιστεύω ότι στην ψηφοφορία θα έχουμε στήριξη για την έκθεση όπως έγινε και με την Οπλή Νομικών Υποθέσεων. Ευχαριστούμε, Μπόνι, για την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Και σε σας ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ για την έκθεση αυτή που είναι ισορροπημένη, έχει μια ισορροπημένη προσέγγιση. Εμείς την εξετάσαμε από πλευρά της ΛΥΜΠΕ. Χρειαζόμαστε την ψηφιακή εναρμόνιση στην Ευρώπη. Τι σημαίνει τώρα ισορροπημένη προσέγγιση. Σημαίνει ότι δεν έχουμε πετύχει την κρίσιμη καμπή, δηλαδή να πούμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερες λύσεις, εναρμόνιση σε περισσότερους τομείς, ανάλυση του εύρους, την ε, ανάπτυξη στοιχείων και προσόντων. Από την άλλη μεριά όμως πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση και ανοίγουμε το δρόμο για την οδηγία για τον ιδιωτικό βίο και την ισορροπία ανάμεσα στην προστασία του ιδιωτικού βίου και τις ευκαιρίες των επιχειρήσεων. Αυτό δείχνει ότι αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντική είναι η προστασία των δεδομένων στην σημερινή μας οικονομία. Χρειαζόμαστε λοιπόν και στο μέλλον λύσεις. Τώρα μπορούμε να ξέρουμε πώς θα μοιραστούμε τα δεδομένα. Τι σημαίνει ε, το που ανήκουν τα δεδομένα. Χρειάζονται και άλλες λύσεις πάντως όσον αφορά την προστασία των δεδομένων. Ευχαριστώ. Εκ μέρους της Επιτροπής, ο Αντιπρόεδρος Άντσιπ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Αξιότιμε Πρόεδρε, αξιότιμε Ευρωβουλευτέ, κυρίες και κύριοι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την έκθεση δύο πρωτοβουλίες όσον αφορά την ψηφιακή ενιαγορά μας βοηθάει να προχωρήσουμε σε διάφορους τομείς πολύ σημαντικούς για την Ευρώπη. Πρέπει να διασφαλίσουμε για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις ότι μπορούν να επωφεληθούν από μια καλά λειτουργούσα ψηφιακή αγορά. Αυτό αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι επίσης ένας τομέας όπου η Ευρώπη έχει να, πει, έχει να μιλήσει για πολλές επιτυχίες. Όντως με τους συνομοθέτες μπορούμε να συνεργαστούμε και αυτό αποτελεί κλειδί για την επιτυχία μας. Ευχαριστώ λοιπόν τις εισηγήτριες, ευχαριστώ και όλους τους ευρωβουλευτές που συμμετείχαν στην εκπόνηση της έκθεσης αυτής. Η ενιαία ψηφιακή αγορά και σχετική στρατηγική αναφέρεται σε συγκεκριμένα θέματα και πρωτοβουλίες. Στο Δεκέμβριο του 2015 ήδη είχαμε υποβάλει μια ανακοίνωση για το copyright με νομοθετική πρόταση όσον αφορά τη διασυνοριακή διάσταση. Αυτό σημαίνει ότι θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι όσοι είναι γεγραμμένοι για διασυνοριακές υπηρεσίες θα παίρνουν αυτό για το οποίο έχουν πληρώσει, ακόμη και αν βρίσκονται σε άλλη χώρα από εκεί όπου αυτό πωλείται. Η επικοινωνία πάντως είναι πολύ βασικό. Έχουμε θέσει στόχους με συγκεκριμένα μέτρα και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Έχουμε υποβάλει μάλιστα και νέα νομοθετική ρύθμιση για την προστασία των καταναλωτών που αγοράζουν ψηφιακό περιεχόμενο ή αγαθά online οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θέλουμε να βοηθήσουμε και τις επιχειρήσεις να επεκτείνουν τις πωλήσει τους online. Όπως βλέπετε, Ήδη προσφέρουμε αποτελέσματα στα πλαίσια αυτής της ενιαίας ψηφιακής αγοράς και θα συνεχίσουμε και το 2016. Επιπλέον, πέρα από τις λύσεις που προτείνουμε για το γεωγραφικό αποκλεισμό, εντοπίζουμε και το θέμα των πληρωμών για τις επιχειρήσεις και όλους τους εμπλεκόμενους. Ο γεωγραφικός αποκλεισμός αντιβαίνει με την ίδια την ιδέα της ενιαίας αγοράς χωρίς σύνορα. Γιατί δημιουργεί ακριβώ σύνορα ανάλογα με την χώρα προέλευσης ή κατοικίας. Οι καταναλωτέ οι επιχειρήσεις startups, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θέλουν να στηρίξουν τον ευρωπαϊκό κλάδο μέσω της ψηφιακής μεταμόρφωσης. Αυτό θα βοηθήσει και για περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Ο κλάδο αυτό είναι πολύ βασικό για την ευρωπαϊκή οικονομία, ο ψηφιακό δηλαδή. Πρέπει να επικεντρωθούμε επίση και στα προσόντα και τι δεξιοτεχνίε του εργατικού προσωπικού. Τον επόμενο μήνα θα κοιτάξουμε και τους κανόνες που ισχύουν για τις τηλεπικοινωνίες και για τα ψηφιακά και τον ιδιωτικό βίο. Ο κυβερνοχώρος, οι δραστηριότητες στο cloud, το λεγόμενο. πώς θα έχουμε εύκολη διακίνηση δεδομένων. Προσβλέπω λοιπόν στις δικές σας απόψεις κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που θα έχουμε και σε συνεργασία μαζί σας, ώστε η ψηφιακή ενιαία αγορά να αποτελέσει πραγματικότητα και ιστορική καμπή για την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε και τώρα από τις πολιτικές ομάδες. Από το ΕΛΚ Βίρκουνεν για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω και εγώ να ευχαριστώ τις εισηγήτριες και τις ε, επιτροπές που έχουν συνεργαστεί ε, στην υπόθεση αυτή βεβαίως και θέλουμε να προχωρήσει το χετεροδυνατό αυτή η ψηφιακή εσωτερική αγορά είναι απαραίτητη για την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη της θέσης εργασίας. Δυστυχώς υστερούμε πολύ σε σχέση με την Ασία και τη Βόρεια Αμερική. Πρέπει λοιπόν αυτές οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες να παρέχονται με τους ίδιους όρους όπως και οι παραδοσιακές διάφτες. Τα ηλεκτρονικά βιβλία, παραδείγματι, θα πρέπει να φορολογούνται όπως και τα κλασικά βιβλία επί Θα πρέπει να έχουμε κανόνες ωστόσο ευέλικτους που θα επιτρέπουν την αξιοποίηση κάθε δυνατότητας που συνεπιφέρει το διαδίκτυο. Χαίρομαι που το Κοινοβούλιο προτείνει την κατάργηση της του περιτού γεωγραφικού αποκλεισμού. Είναι πολύ σημαντικός αυτός για τον χρήστη του διαδικτύου για να μπορεί να αξιοποιεί τις υπηρεσίες, τις διαγραμμικές και έξω από τα εθνικά σύνορα. Έχουμε να κάνουμε μια αγορά 500 εκατομμυρίων κατοίκων και μια εξαίρετη ευκαιρία για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Πρέπει λοιπόν τώρα να πείσουμε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν αυτές ακριβώς τις ευκαιρίες. Οι πολιτικές ομάδες μπορούν να αναπτύξουν τη δική τους γραμμή, αλλά αυτή τη στιγμή είναι κάπως προθύστερο να εφαρμόσουμε την ε, λογική των γαλάζιων καρτών ε, δεν έχει κάποιο νόημα. περιμένουμε τη συνέχεια της συζήτηση για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Η κυρία Κομπούλα Νάτρη. Ε, μία πέτρα παρακαλώ για. Για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι προκλήσεις και τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε σχέση με τις επενδύσεις, την οικονομική ανάπτυξη, τις θέσεις απασχόλησης, οι ελπίδες των νέων, όλα αυτά είναι προβλήματα που θα πρέπει να τα δούμε ως ευκαιρίες και να δράξουμε την κάθε ευκαιρία ε, που προσωποποιεί ουσιαστικά η ενιαία ψηφιακή αγορά. Οι καινοτομίε στι μικρομεσαίε επιχειρήσει είναι μια ευκαιρία για να δημιουργήσουμε θέσει απασχόληση. Η ψηφιακή οικονομία προχωρά πιο γρήγορα από κάθε άλλο τομέα και μπορούμε να δημιουργήσουμε θέσει απασχόληση ποιότητα εδώ. χάρη στην πρόταση της Επιτροπής και τη δική μας έκθεση έχουμε τα θεμέλια για μια δικαιότερη και πιο ολοκληρωμένη ψηφιακή κοινωνία. Υπάρχει ένα ψηφιακό χάσμα το οποίο θα πρέπει να γεφυρώσουμε και στις εγκαταστάσεις ή στις δεξιότητες των πολιτών. Θα πρέπει όλοι οι πολίτες να έχουν πρόσβαση στις ε, υπηρεσίες του διαδικτύου είτε είναι δημόσιες, ε, από δημοσίους δηλαδή παρόχους, είτε είναι ιδιωτικές. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η ε, ψηφιακή ενιαία αγορά δεν θα σημάνει την αρχή νέων κοινωνικών αποκλεισμών. Εκεί θα είναι σημαντική η δική μας ε, η συνεισφορά και θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι υπάρχουν επενδύσεις στα δίκτυα του 5G για να είμαστε βέβαιοι ότι η Ευρώπη έχει την ασφαλέστερη και πλέον προηγμένη δομή και εγκαταστάσεις υποδομές στον κόσμο. Χρειαζόμαστε επίσης στήριξη για την καινοτομία, την ανάπτυξη κρίσιμων υποδομών και ασφαλέστερο κυβερνοχώρο, ασφαλέστερο διαδίκτυο. Χρειάζεται ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για να προωθήσουμε όλους αυτούς τους χώρους και μια ευρωπαϊκή λύση, διότι δεν έχει κανένα νόημα να έχουμε μια ενιαία αγορά ψηφιακέ υπηρεσίε, εάν λειτουργούν εντό των συνόρων μιας και μόνο χώρα. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η προστιθέμενη αξία της ψηφιακή ενιαία αγορά είναι κάτι που θα ωφελήσει όλου του πολίτε. Πρέπει να επενδύσουμε στις υψηλή ταχύτητα υπηρεσίε και να αναπτύξουμε νέα καινοτόμα προϊόντα. Εάν θέλουμε να πετύχουμε και αν τα καταφέρει αυτός ο κλάδος της οικονομίας μας ε, θα γίνει μόνο υπό τον όρο ότι ψηφιοποιείται αλλιώ θα μετεγκατασταθεί αλλού. Το ίδιο και με την αλυσίδα τεχνολογικών λύσεων. Πάντως, η ψηφιακή ένωση πιο πολύ αφορά τις αλλαγές σε κοινωνικό επίπεδο. Κάτι που απαιτεί πολιτική βούληση και ηγεσία. Για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες είναι πολύ σημαντικό η ε, ψηφιακή ενιαία αγορά να προσφέρει νέες ευκαιρίες ας την απασχόληση, τις υπηρεσίες, την ανάπτυξη των απόκεντρων περιοχών και ούτω καθεξής. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει σε συνεργασία με την υπόλοιπη κοινωνία. Ευχαριστούμε Ε, των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών, η κυρία Φόρντ. Σας ευχαριστώ. Εάν θέλουμε να πετύχουμε σε αυτόν τον κόσμο τον ανταγωνιστικό, πρέπει να φροντίσουμε για νέες ευκαιρίες και πλατφόρμες οι οποίες να επιτρέπουν την οικονομική ανάπτυξη και να μπορέσουμε συγχρόνως να αντιμετωπίσουμε προβλήματα της κοινωνίας. Ναι, υπάρχουν αλλαγές. Υπάρχουν διακρίσεις ανάμεσα σε επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, τις αγορές. Σίγουρα υπάρχουν αλλαγές, συνεχείς αλλαγές που οδηγούν και σε νέες προκλήσεις. Όμως πάνω απ' όλα πρέπει να ενισχυθεί η ψηφιακή οικονομία, όχι να υπονομευθεί. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους, να μην εμποδίσουμε την κοινοτομία και τους καινοτόμους και να μην προσθέσουμε κόστος. Η έκθεση αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ακριβώς αυτό το θετικό τόνο χρησιμοποιεί τελευταίες δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η πρότασή της για τις ψηφιακές αγορές, οι διαφορές online, offline, δεν μπορώ να πω ότι είναι αποτελεσματικές όσο θα θέλαμε και όπως επίσης και η αντιμετώπιση των κινδύνων δεν είναι αποτελεσματική από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χρειαζόμαστε σαφείς κανόνους, χρειαζόμαστε συγκεκριμένα στοιχεία για το ωφέλη που έχουμε από το ψηφιακό αυτό περιεχόμενο. Γνωρίζω ότι οι διαπραγματεύσεις τη τελευταίες στιγμή δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για να πετύχουμε ε, σαφή νομοθεσία με συνοχή. Η ενιαία αγορά ε, είναι σε 28 χώρες μέλη που θέλουν να μπορούν online να έχουν δραστηριότητες. Άρα πρέπει να συνεργαστούμε όλοι, σε ολόκληρη την Ευρώπη, για να είναι σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο προστατευτισμός δεν βοηθάει. Ευχαριστούμε. Καράντσοβα. Τώρα, δύο λεπτά παρακαλώ. Εκ μέρους της ομάδας των φιλελεύθερων, Άλτε. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, όπως έγινε και με τη βιομηχανική επανάσταση που μας ε, κατέστησε ηγέτες παγκοσμίω, έτσι και τώρα η ψηφιακή αγορά μπορεί να προσφέρει ανάπτυξη και θέσεις απασχόληση. Η ψηφιακή επανάσταση είναι η νέα βιομηχανική επανάσταση για μα. Όπως και τότε υπήρχαν πολλοί άγνωστοι και φόβος, έτσι και τώρα υπάρχει τάση για προστατευτισμό και φόβος απέναντι σε νέα καινοτόμα μοντέλα. Όμως αυτά ακριβώ θα βοηθήσουν. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι θα προσαρμοστούν και αυτοί που θα μείνουν πίσω. Σήμερα λοιπόν, αν θέλουμε να συνεχίσουμε με τα ίδια επίπεδα ζωής, εμείς ως κοινωνία πρέπει να υποστηρίξουμε την ψηφιακή επανάσταση, η οποία λαμβάνει χώρα έτσι κι αλλιώς γύρω μας. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε και εμείς τα σωστά βήματα για να δημιουργήσουμε μια πραγματική ψηφιακή ενιαία αγορά, να υποστηρίξουμε πολιτικές όπου η καινοτομία και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα, τα νέα προϊόντα, οι νέες αλυσίδες προμήθειας είναι κάτι που θέλουμε. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι πλατφόρμες και η επιμερισμένη οικονομία δεν θα εμποδίσουν την οικονομική μας ανάπτυξη. Αντίθετα, θα αποτελέσουν τον μοχλό της. Ο προστατευτισμός είναι κάτι ξεπερασμένο όσον αφορά την ψηφιακή αγορά. Κύριε Επίτροπε, Στη στρατηγική σας για την ενιαία ψηφιακή αγορά ε, έχετε θέσει 16 ζητήματα υπέρ της ψηφιακής αυτής επανάστασης. Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι έχετε τη στήριξη της ομάδας ALDE για να τα καταφέρετε. Πρέπει να εφαρμόσουμε τη στρατηγική αυτή ολόκληρη γιατί τελειώς η Ευρώπη θα μείνει πίσω. Το αν θα πετύχουμε ή θα αποτύχουμε εξαρτάται αποκλειστικά από εμάς και εμείς μπορούμε να δράσουμε τώρα. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αύριο θα επιβεβαιώσουμε με την ψήφο μας την πολιτική εντολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να χρησιμοποιήσει όλες τις, δυνάμει δυνάμεις προς αυτή την κατεύθυνση. Κύριε Επίτροπε, χρησιμοποιήστε το πολιτικό σας κεφάλαιο. Έχουμε ήδη καθυστερήσει. Ευχαριστώ. Κυρία Έρνστ, ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τις, ε, τις συνεισηγήτριες για την έντιμη συνεργασία. Πρέπει να το σημειώσω αυτό. Δεν ήταν εύκολη η έκθεση. Δεν ξέρω αν μπορούν να αρκέσουν τα σχέδια της Επιτροπής για να εξασφαλίσουν την ταυτόχρονη πρόσβαση στην ψηφιακή εσωτερική αγορά για όλους. Γι αυτό, είναι για, αυτό είναι για μένα ακόμη ακριμές και αυτό πρέπει να επιδιώξουμε με τους αγώνες μας. Έγινε λόγος για τον καταναλωτή, τον πολίτη, τις ανάγκες του. Πολύ σημαντικό, αλλά δεν είναι και αυτονόητο. Εμεί θέλουμε οι καταναλωτές να έχουν την εμπιστοσύνη στα δεδομένα, στην ειλικρίνεια του παρόχου. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό προκειμένου να αναπτυχθεί κατά τρόπο ισοδίκαιο και αποτελεσματικό το διαδίκτυο. Και ξεκινάω από τον δεινόσαυρο που ονομάζεται γεωγραφικός αποκλεισμός. Αυτός πρέπει να πάει στο μουσείο φυσικής ιστορίας, δεν έχει καμία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πρέπει να ισχύει και για το υλικό, το περιεχόμενο που αφορά ε, μειονότητες και για τηλεόραση. Επίσης, το ελεύθερο ε, λογισμικό, το free software, πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο. και βέβαια αυτό προς όφελος του καταναλωτή με αυστηρότερους ελέγχους. Επίσης, η απλούστευση των όρων, κυρίως για τους μικρότερους, όχι μόνο για τους μεγαλύτερους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ εξ ονόματος των Πρασίνων Ρέντα Τζούλια. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Η Επιτροπή έχει ονομάσει την, ε, το εγχείρημα αυτό ψηφιακή εσωτερική αγορά, αλλά δεν πρέπει να λησμονούμε τη σημασία της ανταλλαγής ε, πληροφοριών δεδομένων υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι να χειραφετήσει και να δώσει δύναμη στον πολίτη για την Ευρώπη και για ολόκληρο τον κόσμο, όχι για ορισμένους εκλεκτούς. Δεν μπορούν λοιπόν μόνο οι κερδοσκοπικές επιχειρήσεις να ε, απομιζούν το κέρδος, το όφελος από αυτό το, την ιστορική αγορά. Χρειάζεται ένα λειτουργικό το οποίο θα είναι χρήσιμο, αξιόπιστο. Χρειάζονται υπηρεσίες προς και τις πιο απομακρυσμένες ε, περιοχές. Χρειάζονται επιχειρήσεις ε, με το σύστημα του crowdfunding που θα μπορούν να σταθούν απέναντι στις ισχυρές κεφαλαία και επιχειρήσεις. Χρειάζονται δηλαδή αρκετές αλλαγές ώστε οι νέες τεχνολογίες και οι νέες επιχειρησιακές μέθοδοι να λειτουργήσουν κατά τρόπο αξιόπιστο, χωρίς όμως να χρειάζεται και να επανεφευρεθεί ο τροχός ως προς τον διαμεσολαβητή της υπηρεσίας. Έχουμε να κάνουμε με μια ψηφιακή αγορά που ξεπερνά τους όρους ενός απλού εμπορικού κέντρου. Χρειάζεται συνεργασία, χρειάζεται συμπλήρωση από μια κοινή ψηφιακή στρατηγική προς την οποία τίνει και αυτή η έκθεση. Γι' αυτό και ευχαριστώ τις εισηγήτριες για την πολύ καλή δουλειά και την πολύ καλή συνεργασία στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ. Η FDD Μπορέλη. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η έκθεση αυτή ουσιαστικά μας προϊονίζει μια σειρά από νομοθετικές προτάσεις που θα φτάσουν φέτος στα χέρια μας. Θα μπορούσαμε να είμαστε όμως πολύ πιο φιλόδοξοι, διότι στην υλοποίηση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς ε, η ε, περίπτωση του πολίτη είναι αυτή που θα πρέπει να έχει κεντρικό ρόλο. Ε, Εμεί είμαστε το μόνο θεσμικό οργανό που έχουν άμεσα εκλέξει πολίτε και έχουμε ευθύνη απέναντί του. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να το αποφασίσουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Οι τρει ανακοινώσει που έχουν προαναγγελθεί ω ε, σημαντικότερε στην ιστόση αυτή τη στρατηγική, μα μας υποχρεώνουν να είμαστε ε, πιο φιλόδοξοι και να κάνουμε περισσότερη δουλειά σε σχέση με την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακόμη και για την πώληση εμπορευμάτων στο διαδίκτυο. Δεν έχει αναπτυχθεί πλήρω αυτό ο τομέα στην Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση. 14% μόνο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων τη Ευρώπη χρησιμοποιούν ε, την, ε, το διαδίκτυο για να πολλούν. Πρέπει λοιπόν και οι πολίτε και οι εταιρείε να μπορούν να αγοράσουν και να πουλήσουν ε, στο διαδίκτυο με περισσότερη εμπιστοσύνη και λιγότερα προβλήματα. Δεν πρέπει να υπάρχουν φραγμοί για τι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει, Πρέπει να το ξεπεράσουμε και να υπερβούμε αυτό το φραγμό για να δημιουργηθούν περισσότερες θέσει απασχόληση. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε Τροστίνσκι από την Ευρώπη των Εθνών της Ελευθερίας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όλοι συμφωνούμε ότι οι ψηφιακέ εξελίξει προσφέρουν στι μικρομεσαίε επιχειρήσει δυνατότητε ανάπτυξη. Και αν μπορούμε να βελτιώσουμε το οικονομικό πλαίσιο για αυτέ, θα πούμε ναι. Όμω έχετε πάρει λάθο δρόμο, προσπαθώντα για άλλη μια φορά να σβήσετε τα εθνικά συμφέροντα, ε, ενώνοντα και ενοποιώντα την ψηφιακή αγορά και ξεχνώντα ότι η ευημερία των Ευρωπαίων και ιδίω των Γάλλων ε, θα οδηγήσει σε απορρίθμιση θα, ε, δεν θα ωφεληθεί από την απορρίθμιση των υπηρεσιών που θα οργανωθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για τους χρήστες και για τους παρόχους το ίδιο. Όλα αυτά λοιπόν ε, ε, μας οδηγούν να θέλουμε να καταψηφίσουμε στην ψηφοφορία την έκθεση αυτή. Ναι λοιπόν στις υπηρεσίες, ναι στο όφελος του καταναλωτή, ναι στην διοργάνωση και τη διεντολογία στο διαδίκτυο, αλλά όχι στην ομοσπονδιακή ε, ομοιρία και την ε, προώθηση των διακρατικών οικονομικών συμφερόντων. Συνεργασία των εθνών και όχι διάλυση και καταπαράθρωση αυτών θέλουμε στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε για τους μη εγγεγραμμένους Κόρβιν Μίκε για ένα λεπτό. Ε, ευχαριστώ. Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς συμβαίνει. Μιλάμε για μια αγορά. Εδώ προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια ψηφιακή ενιαία αγορά για να συμπληρώσουμε την εσωτερική μας αγορά. Μα αυτό είναι ένα κλασικό παράδειγμα της τρέβλωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί θα οδηγήσει στην απελευθέρωση των γυναικών. Αυτό είναι κάτι πραγματικά άσχετο, γιατί δεν βλέπετε ποιος είναι από πίσω όταν βρίσκεστε στο διαδίκτυο με ποιον συνομιλείτε. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Ξεκινάει η συζήτηση με τον κύριο Σφάμπ για 1,5 λεπτό. Παρακαλώ. Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, βεβαίω και εγώ εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο θέλω να ευχαριστώ όλου του συναδέλφου που συνέβαλαν σε αυτή την πολύ καλή ε, έκθεση και που πιστεύω θα μπορέσει να εγκριθεί συνενετικά τα λέω μετά τη συζήτηση. Υπάρχει μία προσέγγιση σχετική με την ψηφιακή ιστορική αγορά που μπορεί να έχει ε, αντίκτυπο σε κάθε τομέα της πολιτικής. Γι' αυτό εμείς ως Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θελήσαμε στο πλαίσιο αυτής της εκθέσεως να βρουν τη θέση τους όλες οι επιτροπές. Και ιδιαίτερα έγιναν δεκτές τροπολογίες οι οποίες διεύρυναν το φάσμα της ε, έκθεσης. Κατά τρόπον ώστε όμως να είναι αποδεκτές και για όλους τους εμπλεκόμενους. Το Big Data παραδείγματι. Ήδη το εξέθεσε ο συναρφός Μπόνι. Χρειάζεται μια πραγματική ψηφιακή αγορά για τον καταναλωτή, πέραν των συνόρων, για τον καταναλωτή όπως και για τον εργαζόμενο όμως. 1,5 λεπτό, λεπτό είχα πρόεδρε, μπορώ να συνεχίσω. Ευχαριστώ. Ε, και επίσης φορολογικό δίκαιο, εργατικό δίκαιο και βέβαια τι σημαίνει καινοτομία. Και εδώ θέλω να δώσω την απάντηση ότι καινοτομία είναι και disruption διακοπή, αλλαγή συμπεριφοράς. Αλλά το disruption μόνο του, η διατάραξη δεν αποτελεί καινοτομία. Και βεβαίως εδώ πρέπει να καταπολεμηθεί το ε, geo-blocking, ο γεωγραφικός ε, αποκλεισμός, είναι πάρα πολύ σημαντικό και η εκθέση ήταν πολύ καλή. Ευχαριστώ πρόεδρος. Με συγχωρείτε κύριε Σουάπ, ε, που σας διέκοψα πριν με το σφυρί μου. Είχα μόλις καθίστες του Προέδρου και έκανα λάθος στον κατάλογο και στον χρόνο των ομιλητών. Κύριος Νίκα. Προκειμένου να έχουμε μια πραγματικά ολοκληρωμένη ψηφιακή αγορά, απαιτούνται επενδύσεις στις υποδομές και στα δίκτυα. Και γρήγορα μάλιστα, πάρα πολύ γρήγορα, ακόμα και στην Ήπεθρο, στις απομακρυσμένες περιοχές. Στηρίζω λοιπόν το, τις προσπάθειές μας όσον αφορά τον αδικαιολόγητο γεωγραφικό αποκλεισμό, προκειμένου να υπάρχει εύκολη πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο να μην υπάρχουν επίσης ούτε διακρίσεις όσον αφορά τις τιμές εξαιτίας της ε, γεωγραφικής διάστασης. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής βοηθάει την ε, μεταφορά και την λειτουργικότητα υπέρ του περιεχομένου και των υπηρεσιών που αγοράζονται βέβαια νόμιμα. Πρόκειται επίσης για την πρόσβαση και για την καλή λειτουργία διασυνοριακά Είμαι υπέρ της εδαφικότητας και των μέτρων που καταργούν τους φραγμούς στην ε, μεταφορά περιεχομένου. Βρισκόμαστε στην αρχή της κατάργησης του γεωγραφικού αποκλεισμού. Ευχαριστώ. Henkel. Κυρίες και κύριοι, πριν να εμπλακώ με την πολιτική πριν από δύο χρόνια, ήμουν επί 25 ετία και με την IBM κυρίως της Γερμανίας δραστήριο στον τομέα αυτό. Είχα επαφές και με συνδικάτα και με ε, κλησιαστικές οργανώσεις και με πολιτική και με μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να προστατευτούν οι πολίτες από την αυτοεκμετάλλευση. Θα χρειαστεί να επισημάνουμε τα δυσάρεστα αυτής της έκθεσης, έστω και αν πρέπει να τα δεχθούμε. Οι πολίτες θέλανε όλο και περισσότερη συνδιαμόρφωση και λιγότερη αυτοδιάθεση. Θεωρείται. Θεωρείται επίσης ότι αυτή η ιδιωτική πρωτοβουλία μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερη δημιουργικότητα. Ότι δεν χρειάζεται δαιμονία από τις κρατικές δομές. και ότι αυτή μπορεί να πλήξει τις επιχείρησεις μας. Όταν λοιπόν διρωτώμεθα γιατί η ψηφιακή Ευρώπη έχει τέτοια επιτυχία στην, στις ΗΠΑ και την Ασία, η απάντηση είναι ότι δεν, δώσαμε, δεν δείξαμε αρκετή εμπιστοσύνη στις επιχειρήσεις μας και τους πολίτες. Δεν τους δώσαμε αρκετές ελευθερίες. Μόνο με την ελευθερία και την ε, υπευθυνότητα μπορεί να υπάρξει αυτή η δημιουργικότητα και στην ψηφιακή αγορά και θα ήθελα καταλήγοντας να πω έτσι προτέρα κένσο πρέπει να καταργηθεί η εσωτερική αγορά. Ο πρόεδρος. Κυρία Γιάκο Κοσάρη έχει μια ερώτηση. Κύριε Χένκελ, τη δέχεστε. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε. Είπατε ότι η Ευρώπη υστερεί ως προς την ψηφιακή της ανάπτυξη γιατί δεν δόθηκε αρκετή εμπιστοσύνη στον επιχειρηματία και τον πολίτη. Ναι, αλλά η ανάλυση είναι ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα 28 κράτη-μέλη επέλεξαν την προστασία, την εθνική για, την για τα προσωπικά δεδομένα και όλες τις άλλες ε, ψηφιακές αξίες. Μήπως αυτό είναι το οποίο θα πρέπει να κοιτάξουμε ως προς την αξία της εσωτερικής ψηφιακής αγοράς. Κύριε Σφέγκελ, συμφωνώ, έχετε δίκιο ότι ο κατακαιρματισμός της εσωτερικής ψηφιακής αγοράς αποτελεί έναν από τους λόγους, αλλά δεν είναι ο μοναδικός, δεν είναι ο κύριος καν λόγος. Ο κύριος λόγος είναι ότι δόθη εμπιστοσύνη στην κρατική παρέμβαση. Μπορώ να σας δώσω καταλόγους ε, προγραμμάτων υποστήριξης της πολιτικής τεχνολογίας αμέτρητος. Όλες αυτές οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, Νίξτορ, Φολιβέτη, Siemens, Μπούλ, ICL, εξαφανίστηκαν. Οι Αμερικανοί όμως όχι, οι Αμερικανικές όχι. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ όμω να προσέχετε. Στα 30 δευτερόλεπτα θα διακόπτω τον ερωτώντα και στα επόμενα 30 τον απαντώντα. Ε, κυρία Τούμτορ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Οι συνάδελφοι συμφωνούν ότι θέλουμε ψηφιακή αγορά. Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι στη ζωή μας καθημερινά. Δυστυχώς η ευρωπαϊκή νομοθεσία και οι ευρωπαϊκές πολιτικές δεν ανταποκρίνονται στις προκλήσεις και κάποιες χώρες δεν τα καταφέρνουν καλά. Στη δικιά μου χώρα μπορεί κανείς να φτιάξει online μία επιχείρηση μέσα σε μισή ώρα. Και μπορεί να έχει πρόσβαση κανείς σε αυτήν μέσω του διαδικτύου από παντού στον κόσμο. Δεν ισχύει όμως κάτι αντίστοιχο σε όλες τις χώρες μέλη. Τα εμπόδια είναι πολλά. Η ηλεκτρονική υπογραφή είναι κάτι που χρησιμοποιείται ευρέως. Όμως εξακολουθούν να υπάρχουν σύνορα ακόμα και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είναι ένα καυτό ζήτημα αυτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχουν 16 κατευθύνσεις που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προχωρήσουμε με αυτό το θέμα αλλά εξακολουθούμε να πρέπει να αντιμετωπίσουμε βασικά ζητήματα για να λειτουργήσει καλά μια ενιαία ψηφιακή αγορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Τόμ. Ο κύριος Ιλκιώτης. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η ψηφιακή ενιαία αγορά θα επιστρατεύσει δυστυχώ τι νέε τεχνολογίε για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πολυεθνικών και του μεγάλου κεφαλαίου. Αντί πρωταρχικός στόχο να είναι ευημερία και ενίσχυση τη ποιότητα ζωή των ανθρώπων οι δυνατότητε τεχνολογία θα αξιοποιηθούν δυστυχώ κυρίω για την αύξηση των επιχειρηματικών κερδών και τη ανταγωνιστικότητα. οι μεταρρυθμίσει που προωθούνται για ολοκλήρωση τη ενιαία ψηφιακή αγορά θα έχουν ιδιαίτερα αρνητικέ επιπτώσει στι μικρομεσαίε επιχειρήσει στα εργασιακά δικαιώματα αλλά και στου ίδιου του καταναλωτέ. χρειάζεται λοιπόν να επαναπροσδιοριστούν οι στόχοι τη ψηφιακή ατζέντα ώστε στο επίκεντρο να τεθούν τα συμφέροντα τη κοινωνία. η θέση μα είναι ξεκάθαρη η υλοποίηση τη ψηφιακή αγορά πρέπει να συμβάλλει στη δημιουργία νέων ποιοτικών θέσεων εργασία στην ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων αλλά και των δικαιωμάτων των καταναλωτών. εξίσου σημαντικό είναι να διασφαλιστεί η ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο αλλά και η προστασία των προσωπικών δεδομένων. επίση η τεχνολογία πρέπει να αξιοποιηθεί ώστε να ενισχυθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ιδιαίτερα όσον αφορά την πρόσβασή τους στη χρηματοδότηση αλλά και τη θέση τους στην αγορά. προς αυτή την κατεύθυνση είναι και οι τροπολογίες που κατατέθηκαν εκ μέρους της ευρωπαϊκής ενωτικής αριστεράς. ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τάραντ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ως πρόεδρος της Εσθονικής Ένωσης ε, των Ατόμων με Προβλήματα Κινητικότητας και αντιπρόεδρος της, ομάδας, ε, της διαπολιτικής ομάδας ε, για τα άτομα με αναπηρία εδώ στο Κοινοβούλιο. Βλέπουμε ικανοποίηση ότι αναφέρονται και τα άτομα με αναπηρία στην έκθεση και ότι αναφέρεται η δυνατότητα της πρόσβασης και οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, όπως άλλωστε και αυτό της, το πρόβλημα της ενσωμάτωσης στην αγορά εργασίας. Επίσης, πολύ σωστά επισημαίνει η έκθεση το λυπηρό γεγονό ότι η ψηφιακή ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής, Αγοράς, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν ικανοποιεί τις ανάγκες για πλήρη και περιόριστη πρόσβαση και των ατόμων με αναφήρεια στις ε, ε, δυνατότητες ψηφιακής αγοράς, η προσβασιμότητα, η διαλειτουργικότητα. Πρέπει ωστόσο να υπογραμμιστούν περισσότερο στην έκθεση. Θα μπορούσαμε να έχουμε καταπληκτικό λογισμικό για τους τυφλούς και τα άτομα με οπτικές δυσκολίες. Ε, ωστόσο αυτό περιορίζεται μόνο σε ιστοσελίδες, περιεχόμενο κτλ. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει οι ελεύθερες ε, και ομοιόμορφες προδιαγραφές να ισχύουν σε όλη την αγορά. Ε, στην έκθεση, κύριε Επίτροπε, έχουμε 4 με 5 σελίδες κειμένων παράθεση κειμένων ε, ε, που έχουν ήδη εγκριθεί από τους νομοθέτες. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν υλοποιηθεί αυτά που ήδη εγκρίθηκαν στο παρελθόν. Παρακαλώ να με ρημνήσετε στο αυτό να αντιμετωπιστεί. Ο πρόεδρος, ευχαριστώ. Κύριε Τάραντ, δέχεστε μια ερώτηση από τον συνάδελφο Μαλατίτς. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και τις συνεισηγήτριες που μαζί με όλο το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή Συνέταξα να την τόσο ισόρροπη ε, έκθεση. Μα δεν σας έδωσα το λόγο ακόμα. Δεν έχετε το λόγο, ο κύριος Μάλετιτς. Η κυρία Μάλετιτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που δεχτήκατε και τη γαλάζια μου κάρτα. Η Εστονία είναι μία από τις χώρες που έχει ηγετικό ρόλο στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε όλα τα επίπεδα. Θα ήθελα να μου πείτε πώς ε, θα θέλατε να βοηθήσετε άλλα κράτη που είναι λιγότερα προηγμένα, προηγμένα προς αυτή την κατεύθυνση να προχωρήσουν. Ε, τι θα κάνετε για να ενισχύσετε και να μπορέσει να προχωρήσει στην πράξη η ψηφιακή ενιαία αγορά. Σας ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση. Δεν είμαι αρμόδιος να απαντήσω αναγκαστικά. Ο Πρωθυπουργός μας που ήταν ε, υπεύθυνο για τουλάχιστον 9 χρόνια θα μπορούσε να απαντήσει εκείνος. Εγώ ίδιος δεν ξέρω τι να πω ε, για το θέμα αυτό διότι αν ήταν στα δικά μας τα χέρια δεν υπήρχε περιπτώσει να μην έχετε μια πολύ χειροπιαστή απάντηση. Ευχαριστούμε για ένα λεπτό κύριο Τσούλο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και τις συνεισηγήτριες για την δουλειά τους. Η έκθεση αυτή είναι ιδιαίτερα ισορροπή και μπορούμε να την στηρίξουμε. Θεωρώ ε, θεμελιώδες να εντοπίσουμε τρεις πυλώνες ε, στο έργο μας για να μπορέσουν να είναι εφικτά αυτά που ονομάσαμε ψηφιακή ε, γειτονία στο μέλλον. Πρώτα απ' όλα η αρχή της ισότητας, δηλαδή δυνατότητα να έχουμε τα ίδια δικαιώματα για όλους τους χρήστες και να τους τα ε, παρέχουμε είτε στο διαδίκτυο είτε εκτός. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ε, απαλληθούν όλες οι διακρίσεις, κυρίως οι γεωγραφικές. Δεύτερος πυλώνας είναι η συμμετοχή. Νομίζω ότι πρέπει να φροντίσουμε οι πολίτες, ε, οι δημόσιες υπηρεσίες και οι επιχειρήσεις να προχωρήσουν στην ανταλλαγή πληροφοριών και να κάνουν αποτελεσματική αυτή την αγορά. Και μετά πρέπει να επικεντρωθούμε στην εμπιστοσύνη. Θα πρέπει να προβλέψουμε σε αυτή την έκθεση διαφορετικά εργαλεία ώστε ο πολίτης και ο χρήστης να μπορέσουν να προχωρήσουν σε αυτόν τον ε, τομέα. Ε, και θα πρέπει να προβλέψουμε και τα κατάλληλα εργαλεία. Ευχαριστούμε η κυρία Κάπελ. Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ο τομέας της ψηφιακής οικονομίας είναι ένας ε, πολύ σημαντικός τομέας με μεγάλο δυναμικό ε, δυναμικό ανάπτυξης που μπορεί να φέρει και 400 δισεκατομμύρια ευρώ ε, μέχρι και 3,8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Νομίζω ότι πρέπει να πούμε πως η έκθεση είναι πολύ καλή, ισορροπημένη. Αποτελεί μια πολύ καλή βάση εργασίας, καλύπτει πολλά θέματα. Ένα-δύο σημεία μόνο θέλω να επισημάνω. Αυτή η μανία να ρυθμίζουμε τα πάντα, ε, προϋποθέσεις ευθύνης, όροι ε, λειτουργίας, ε, διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία δεν μοιάζουν, δεν μοιάζουν με ρυθμίσεις του 21ου αιώνα. Ας αφήσουμε ανοιχτά ορισμένα ζητήματα πλέον. Και δεύτερον, ανταγωνισμός και επενδύσεις για, την, ε, για τις υποδομές της ευρυζωνικότητας. Ο Πρόεδρος χτυπάει το σφυρί. Ευχαριστώ κυρία Κάπελ. κάρενς ένα μιση λεπτό, μια και ο κύριος Κόβατς δεν είναι εδώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, η ψηφιακή ενιαία αγορά αξίζει το όνομά της. Όλοι εδώ αντιλαμβανόμαστε περί τίνος πρόκειται. Ο κόσμος όμως το καταλαβαίνει. Ας το δούμε πρακτικά. Οποιοςδήποτε από εμά μπορεί να πάει ας πούμε στο Μόναχο να αγοράσει εκεί τα φημισμένα λουκάνικα. Μετά από εκεί μπορώ να πάω στη Ρίγα, στην ε, Στοκχόλμη, στη Λισαβόνα. Είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικό. Συγχρόνως όμως από τη Ρίγα, μπορώ να πληρώσω κάποια συνδρομική για ψηφιακό περιεχόμενο στην τηλεόραση. Δεν μπορώ όμως να το δω ούτε στο Μόναχο, ούτε στο Δουβλίνο, ούτε πουθενά αλλού. Και γιατί? γιατί για τα αγαθά λειτουργεί αυτό καλά. Μπορέσαμε να καταργήσουμε τα σύνορα, ενώ για το ψηφιακό περιεχόμενο που γίνεται όλο και περισσότερο σημαντικό για την ε, οικονομία μας, αυτό παραμένει πάρα πολύ δύσκολο εξαιτία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνία κλπ. κλπ. Λοιπόν, όλα αυτά τα εμπόδια πρέπει να τα καταργήσουμε. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το copyright ισχύει για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα διπλώματα ευρεσιτεχνία. Να μην χρειάζεται να πάμε στο μόναχο για τα περίφημα λουκάνικα, αλλά να μπορούμε από οπουδήποτε να αποφελεθούμε από το διαδίκτυο και το ψηφιακό περιεχόμενο χωρίς εμπόδια. Ευχαριστώ. Κύριε Κάρινς, δέχεστε ερώτηση από τον κύριο Σάνι. Κύριε Κάρινς, δέχεστε ερώτηση από τον κύριο Σάνι. Παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ήθελα να ρωτήσω τους συναδέλφους του ΕΛΚ από πιο πριν εάν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο απαριθμούν τόσα πολλά στοιχεία της ιστορικής ψηφιακής αγοράς που όντως είναι σημαντικά και καλά κάνουν αλλά διερωτώ με μέσα σε όλη αυτή την απαρίθμηση γιατί λησμονείται την εκπαίδευση δεν είναι σημαντικό στοιχείο Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε για την ερώτηση αυτή. Αν ε, μιλάμε για την ε, ενιαία αγορά, στη ψηφιακή ενιαία αγορά από πλευράς του ΕΛΚ, το επιχείρημά μας είναι ότι πρέπει να καταργηθούν τα εμπόδια σε όλους τους τομείς. Όπου υπάρχουν εμπόδια πρέπει να καταργηθούν. Η ψηφιακή εσωτερική αγορά είναι πολύ σημαντική και για την εκπαίδευση και για τα αγαθά και τις υπηρεσίες. Η πολιτική μας ομάδα δηλαδή λέει ότι πρέπει να καταργηθούν όλα τα εμπόδια. Ευχαριστώ ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Μια πλήρως ολοκληρωμένη ψηφιακή αγορά αποτελεί στοιχείο κλειδί της σημερινής Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι ψηφιακές τεχνολογίες προσφέρουν τεράστιες ευκαιρίες. Δημιουργία θέσεων απασχόλησης, δηλαδή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Η ανάπτυξη μπορεί να φτάσει στα 450 δις ευρώ. Οικονομική ανάπτυξη. Όμως υπάρχει πολύ αυστηρή νομοθεσία άκαμπτη στις αγορές τηλεπικοινωνίας της χώρες μέλη και στα θέματα νομοθεσίας copyright πνευματικής διοκτησίας. Άρα χρειάζεται αλλαγή και στη συμπεριφορά των καταναλωτών και χρειάζονται και μεταρρυθμίσεις στη νομοθεσία copyright για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην ψηφιακή επανάσταση. Είναι ζωτική σημασία για την προστασία δεδομένων, προστασία καταναλωτών να έχουμε ενιαίους κανόνες και για να προωθήσουμε την κουλτούρα και την επιχειρηματικότητα. Ευχαριστώ, Ντάλτον, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ψηφιακή επανάσταση είναι εδώ. Θα αλλάξει κάθε τρόπο ζωής, κάθε κομμάτι της καθημερινής μας ζωής, όπως στο παρελθόν η γεωργική και μετά η βιομηχανική επανάσταση. Δεν πρέπει να αναγνωριστεί ότι υπάρχει μια παγκόσμια αγορά που ενώνει Τρία δισεκατομμύρια πολίτες σε όλο τον κόσμο και δεν μιλούμε για μια ευρωπαϊκή αγορά αλλά μια παγκόσμια ψηφιακή αγορά και δεν επιτρέπεται να ορίσουμε ε, φραγμούς. Το, ο γεωγραφικός ε, περιορισμό σε ότι αγοράζουμε κάτι μέσω του διαδικτύου για να μην μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε μετά σε κάποιο άλλο μέρο της γη. Δεν επιτρέπεται αυτό, αλλά ταυτόχρονα δεν πρέπει να υπάρχουν πανευρωπαϊκές άδειε. Ε, θα πρέπει να βοηθήσουμε την sharing economy, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που θέλουν να μοιραίουν την προσπάθειά τους. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε όμως και τις υφιστάμενες επιχειρήσεις. Το διαδίκτυο είναι εξορισμού παγκόσμιο. Είτε πρόκειται για ασφάλεια του νεφούς, του ψηφιακού νεφούς, είτε πρόκειται για το γεωγραφικό αποκλεισμό, είτε πρόκειται για οτιδήποτε άλλο, έρχεται ένα ψηφιακό τσουνάμι και πρέπει να πάμε με το κύμα. Ευχαριστώ πολύ. ένα λεπτό. Ευχαριστώ και επιτρέψτε μου να ευχαριστώ πρώτα τους δύο τις δύο για την πολύ καλή δουλειά τους σε αυτό το σημαντικό θέμα. Έχουμε όλο και πιο πολλά προβλήματα όσο ενισχύεται, όσο αυξάνεται η χρήση του διαδικτύου, η προστασία των δεδομένων, των πληροφοριών, η προστασία η δική μας, ε, χωρίς παραβίαση των, ε, είτε της ελευθερίας, των όρων της ελευθερίας του λόγου ή των προσωπικών μας δεδομένων πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε και τον ιδιωτικό βίο και ένα απαραίτητο επίπεδο ασφάλειας. Χρειάζεται, όπως λέει και η έκθεση, να αποτραπεί η λογοκρισία, η υποβάθμιση της ελευθερίας της έκφρασης μέσω του διαδικτύου λόγω μιας ε, υποχρέωσης, ε, μιας ευθύνης του μεσολαβητή. Πρέπει να υπάρξει έλεγχος του παράνομου περιεχομένου. Δεν μπορούν διαφορές πλατφόρμες να υποκαθιστούν τις αρχές επιβολής του νόμου και της τάξης. Και πρέπει να θυμόμαστε επίσης ότι μιλάμε για την ψηφιακή αγορά της Ευρώπης, αλλά ταυτόχρονα μιλάμε για μια διαγραμμική συμπεριφορά και επικοινωνία που δεν περιορίζεται στα σύνορα της Ευρώπης. Και γι' αυτό πρέπει να έχουμε ασφαλή μετάδοση προσωπικών δεδομένων και σε αυτό καταλήγω ότι χρειάζεται κατεπηγόντως συμφωνία, όχι μόνο με τους Αμερικανούς για το θέμα αυτό, για να υπάρξει ασφάλεια δικαίου για τον Ευρωπαίο πολίτη, για τον Ευρωπαίο καταναλωτή και την Ευρωπαϊκή επιχείρηση. Ευχαριστώ πολύ για ένα λεπτά, λεπτό συνάδελφος Στάλκα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως ακούσαμε, το διαδίκτυο είναι ο κατεξοχήν τρόπος επικοινωνίας της μέρες μας. Υπάρχουν παρόλα αυτά μια σειρά από Και η ομάδα μου, η Ενωτική Αριστερά, στηρίζει την ψηφιακή ενιαία αγορά, όμως πρέπει να επισημάνουμε κάποιες από τις δυσκολίες που πρέπει να υπερβούμε προκειμένου να πετύχει. Λόγω χάρη προστασία των δεδομένων, η προστασία των καταναλωτών, όταν αγοράζουν αγαθά εντός αυτής της ενιαίας αγοράς ή έχουν να κάνουν με τις δημόσιες υπηρεσίες στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, το e-government. Επίσης κάποιοι εργάζονται από το σπίτι τους και εκείνων τα δικαιώματα πρέπει να γίνονται σεβαστά. Η ψηφιακή ενιαία αγορά πρέπει να έχει ένα κεντρικό ε, ρόλο προστασίας. Ευχαριστούμε κύριε Μαστάλκα. Ο κύριος Ρέιμον. Πρόεδρε, Επιτρέψτε μου να επισημάνω κάτι καινούριο σε αυτήν την προχωρημένη ώρα της συζήτηση, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε συζήτηση μόνο για την εσωτερική αγορά. Έχουμε να κάνουμε τα δικαιώματά μας ως καταναλωτών βεβαίω, αλλά ταυτόχρονα και με τα δικαιώματα του πολίτη. Στο γεωγραφικό αποκλεισμό λοιπόν η συζήτηση για το αν ένα Ευρωπαίος μπορεί να δει περιεχόμενο έξω από τη χώρα στην οποία διαμένει. Και αυτό δεν μπορεί να είναι μόνο ένα οικονομικό ζήτημα, δεν μπορεί να είναι ένα ζήτημα καταναλωτή μόνο. Είναι ζήτημα λογοκρισίας. Εάν μπορώ στην Ευρώπη, οπουδήποτε και αν βρίσκομαι, να βλέπω, να διαβάζω, να ακούω ε, οποιοδήποτε περιεχόμενο διαλέξω. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ο κόσμος στο μέσο μαζικής ενημέρωσης έχει αλλάξει. δεν είναι πια αυτός ε, ο, της παραγωγής ε, περιεχομένου για την αναζήτηση μετά του καταναλωτή. Τώρα έχουμε να κάνουμε με μια διαφορετική υποδοχή των δεδομένων και αυτό πρέπει να συζητηθεί με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Ευχαριστώ κύριε Ραϊμόν. Κυρία Πάρκερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η συζήτηση και η ψηφοφορία τη σημερινή συζήτηση είναι χάσιμο χρόνο για το Κοινοβούλιο. Όχι μόνο γιατί διαφωνώ με πολλέ πτυχέ όσον αφορά τη δημιουργία τη ενιαία ψηφιακή αγορά, αλλά και επειδή πριν καν φτάσουμε στην ψηφοφορία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δουλεύει κρυφά για να προχωρήσει η νομοθεσία και να πετύχει έτσι του δικού τη στόχου. Τέτοια βιασύνη όμω δεν είναι υπέρ των καταναλωτών, υπέρ των επιχειρήσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση που θα έχουν να κάνουν ε, με μια κακή νομοθεσία. Το θέμα της πώληση ψηφιακών υπηρεσιών, για παράδειγμα. Όλα αυτά τα κάνουν ε, οι γραφειοκράτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που λίγα ξέρουν από επιχειρήσει. Η πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει αναγκάσει έτσι κι αλλιώς πολλές επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση να διγραμμιστούν με την ενία αυτή η αγορά. Η έκθεση αυτή λοιπόν τολμάει να λέει ότι μέχρι τώρα είχαμε επιτυχίε σε αυτό το τομέα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως δεν τα έχει καταφέρει. Τα επίπεδα είναι πολύ χαμηλά και είναι τροπή να λέμε ότι πρόκειται για επιτυχία. Οι online πωλήσει μάλλον περισσότερα προβλήματα θα δημιουργήσουν παρά θα λύσουν. Ευχαριστώ. Φερχάιεν. 1,5 λεπτό. Είναι πολύ σημαντικό για την οικονομική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό το θέμα και έχει τεράστιο δυναμικό για την ανάπτυξη και πολιτιστικού περιεχομένου και τη διάδοση επιστημονικής γνώσης. Θα πρέπει να εξαντληθούν όλες του οι δυνατότητες έτσι ώστε να μπορέσουμε να διευρύνουμε τον πολιτισμό στην Ευρώπη, να οικοδομήσουμε μια Ευρώπη της γνώσης και να καταστήσουμε και για το μέλλον ανταγωνιστική την ευρωπαϊκή κοινωνία. Χρειάζεται λοιπόν να αναπτυχθούν όλες οι δομές και από μικρούς και μεγάλους παράγοντες της αγοράς. Είναι μεγάλες οι αλλαγές στο ψηφιακό περιβάλλον. Πρέπει να γίνουν όλες αυτές έτσι ώστε στον τομέα των οπτικοακουστικών να γίνει η ε, να καλυφθεί το χάσμα μεταξύ ε, διαγραμμικών και μη διαγραμμικών ε, περιεχομένων και πρέπει ο κάθε ένας από τους παράγοντες να κοιτάξει να αποτρέψει τη τρεφλός στην αγορά. Η Επιτροπή του Πολιτισμού υπογραμμίζει στην έκθεσή τη ότι το οπτικοακουστικό περιεχόμενο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα πρέπει να εισαχθούν ε, προϋποθέσεις για την προστασία της ε, πολυφωνίας και της ελεύθερης έκφρασης. Για τους νέους επίσης θα πρέπει να έχουμε ε, μια ισορροπημένη τοποθέτηση. Η ψηφιακή εσωτερική αγορά με τη στρατηγική της θα πρέπει να καταργήσει τα εμπόδια και να προστατεύσει τον καταναλωτή. Πρέπει να υπάρχει μεταβιβασιμότητα με νόμιμη πρόσβαση σε περιεχόμενο οι οικονομικές όμως συνθήκες πλησίου για την επαγγελματική παραγωγή οπτικοακουστικού περιεχομένου δεν μπορούν να διαταραχθούν και θα πρέπει σε σχέση με τον... Ευχαριστώ πολύ λέει ο πρόεδρος που διακόπτει και ο κύριος Στοσενόφσκι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι ως σκιώδης εισηγητής για την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών αγωνίστηκα και συνεισέφερα και ε, προς την κατεύθυνση της ψηφιακής αγοράς με δική μου έκθεση. Η ενιαία ψηφιακή αγορά δίνει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, τη δυνατότητα να έρθουν σε ανταγωνισμό με πολύ μεγάλες εταιρείες και ομίλους. Είναι πολύ σημαντικό βήμα αυτό για τους νέους Ρουμάνους επιχειρηματίες και υπάρχει πολύ μεγάλο δυναμικό όχι μόνο στη Ρουμανία. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα προσωπικά δεδομένα, το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και την οικογενειακή. Όλα αυτά θα πρέπει να έχουν στο κέντρο τον πολίτη και τη δυνατότητα να ελέγχει τα δεδομένα του. Οι κυρώσεις θα πρέπει να είναι δρακόντιες για να μην γίνονται καταχρήσεις και παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων. Και όταν αυτά διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες θα πρέπει να ελέγχεται αυστηρά η διαδικασία. Η εσωτερική αγορά έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες αλλά μπορεί να μείνει και νεκρό γράμμα ή να διαστρεβλωθεί και να κάνει ζημιά. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ κύριε Τωσενόφσκι. Επιτρέπετε ερώτηση του κυρίου Μπονάνο. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον συνάδελφό μου, τον κύριο Πάβελ, όταν μιλάει για δρακόντιες κυρώσεις, τι ακριβώς εννοεί. Τι έχει υπόψη του, δηλαδή, να επιβάλλεται ως κύρωση εις βάρος κάποιου που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για εγκληματικούς σκοπούς. Λέγομαι Εμίλιαν Πάβελ κύριε Πρόεδρε και σας διορθώνω δεν λέγομαι το Ζενόφσκι ε, και απαντώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στο συναδελφό που μου κάνει την ερώτηση αυτή. Θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι όσοι διαχειρίζονται αυτά τα δεδομένα θα είναι πάρα πολύ ε, τυπικοί και νόμιμοι στη δράση τους. Και όταν υπάρχουν εγκληματικές ενέργειες αυτές να τιμωρούνται. Είμαι βέβαιο ότι υπάρχει δυνατότητα αυτό να γίνει και έχει και συμφέρον ο ιδιωτικό τομέα και τα κράτη-μέλη να προστατεύουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών τους. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πάβελ. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Ε, έδωσα το λόγο στον κύριο Τοσενόφσκι, μου είχε διαφύγει το δικό σας όνομα και νόμιζα ότι είχε μιλήσει και ο κύριος Τοσενόφσκι. Το λόγο είχε ο κύριος Πάβελ, λέει ο πρόεδρος. Μα όχι, τώρα είμαι εγώ, Τοσενόφσκι. Ναι, δεν πειράζει. Να. Κύριος Τοσενόφσκι. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, ακούστηκε προηγουμένως ε, ότι η ψηφιακή αγορά είναι πάρα πολύ σημαντική για ε, την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη και ευημερία. Είναι βασικός ε, στόχος σήμερα, γι' αυτό θα πρέπει να παραμένουμε ενεργοί και δραστήριοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να βοηθούμε όσο γίνεται την ενιαία ψηφιακή αγορά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους για τις προσπάθειες που κατέβαλαν όλες τις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Νομίζω ότι καταφέραμε να δώσουμε Στου έμφαση στους σημαντικούς τομείς για την περαιτέρω ανάπτυξη της ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Το μόνο ερώτημα που παραμένει είναι πώς θα εναρμονιστούν τα τέλη και οι τιμές και η φορολογία που μπορεί ενδεχομένως να είναι σοβαρό πρόβλημα. Εμείς θα πρέπει να υπερασπιστούμε την αγορά απέναντι σε οποιασδήποτε απόπειρες υπερβολικής ρύθμισης να βοηθήσουμε την κάλυψη, την ασφάλεια και την ταχύτητα της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και μέχρι εκεί. Υπάρχει πολύ μεγάλο δυναμικό εδώ για τον ιδιωτικό τομέα ε, που ε, προωθεί τον κλάδο και τον ε, συντηρεί. Γι' αυτό θα πρέπει να ρίχνουμε όλα τα εμπόδια και τους φραγμούς. Ευχαριστώ πολύ για ένα λεπτό η κυρία Σχάκε. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, έχουμε καταθέσει ένα φιλόδοξο κατάλογο επιθυμιών για να περάσουμε το ταχύτερο δυνατόν στην ενιαία ψηφική αγορά ή αν θέλετε στον ενιαίο ψηφιακό χώρο στην Ευρώπη. Ιδιαίτερα αυτούς του ε, χαλεπούς καιρούς ε, πρέπει να προσφέρουμε ελπίδα για καινοτομία, για ε, τεχνολογία και οικονομία της γνώσης. Αυτό είναι καθοριστική σημασία για τις νεοφυείς επιχειρήσεις για να μην φύγουν και αυτέ, να πάνε όλοι στο Silicon βάλει. Χρειαζόμαστε λοιπόν πρακτικές λύσεις για να εναρμονίσουμε τη διαφορετική νομοθεσία για το δικαίωμα του δημιουργού, το copyright και πολλά σύναφη. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον θεμητό ανταγωνισμό και αυτά να παραμείνουν παρά την τεχνολογική επανάσταση. Το ανοιχτό διαδίκτυο, η πρόσβαση, η ουδετερότητα του διαδικτύου, ναι, απαραίτητα, αλλά όχι η ιδιωτικοποίηση ε, στον τομέα της ε, νομοθεσίας. Αυτά είναι πολύ σημαντικά για όλους ανά τον κόσμο, άρα δηλαδή πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στην διαχείριση του ε, διαδικτύου, να μην επιτρέπουμε να υπάρχει έλλειψη ελέγχου. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Χέλμαρ για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν κάποια στοιχεία σε αυτή την πρόταση που θα είναι πολύ δημοφιλή ε, στους ε, ε, εκλογείς. Θα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη να μπούμε στο BBC Plus Service όταν θα είμαι στο Στρασβούργο της Βρυξέλλης. Όμως καταραίουν άλλες ρυθμίσεις για το copyright που έχουμε κάνει. Πολλές επιχειρήσεις χρειάζονται αυτά τα έσοδα για να παρουσιάζουν το απαιτούμενο περιεχόμενο. Εμείς ανησυχούμε για την άκαμπτη νομοθετική δράση της κοινότητα, της Κομισιόν είναι εις βάρος της καινοτομίας και δεν καλύπτει τις ανάγκες των κρατών μελών. Βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός πέραν των συνόρων για να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα του διαδικτύου σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πιστεύουμε όμως ότι ο συντονισμός θα επιτυγχάνεται καλύτερα με την συνεργασία ανεξάρτητων κρατών αντί με το να υπάρχει κεντρικός προγραμματισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπω είπαν πολλοί συνάδελφοι, αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε είναι μια ε, παγκόσμια και όχι απλά ευρωπαϊκή λύση. Ευχαριστούμε πολύ κύριε συνάδελφε. Τώρα για 1,5 λεπτό κυρία Ντελκαστήγιο Βέρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Πολλά πράγματα υπόθηκαν ήδη. Εγώ θέλω να εστιάσω την τοποθέτησή μου σε ένα στοιχείο που είναι κρίσιμο για την ψηφιακή οικονομία και την ψηφιακή αγορά, που είναι η μεγάλη κλίμακα, το μεγάλο πλαίσιο που μπορεί να αναπτυχθεί στην Ευρώπη αυτή η οικονομία. Και αυτά είναι τα δεδομένα. Είναι πάρα πολύ κρίσιμα στην ανάπτυξη της ε, ψηφιακής οικονομίας. Η μαζική ανάλυση, το big data, η ανταλλαγή δεδομένων συνιστούν ένα βασικό άξονα και ένα βασικό πυλώνα μέχρι του εξής βαθμού. Οι αναλυτές τώρα των δεδομένων είναι το κατεξοχήν επάγγελμα ε, που ζητούν στον κόσμο σύμφωνα με μια μελέτη που εκδόθηκε πριν από λίγες εβδομάδες στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Υπό την έννοια αυτή λοιπόν και με αυτά τα δεδομένα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και την διαβίβαση των δεδομένων. Πώς διαβιβάζονται, πώς κυκλοφορούν, γιατί κυκλοφορούν. Υπάρχουν κάποια δίκτυα τα οποία δίκτυα αυτά συνιστούν την υποδομή της ψηφιακής οικονομίας. Παλιά οι μεταφορές ήταν διαξηράς θαλάσσης και αέρος και στην, η οικονομία αυτή την ψηφιακή είναι μέσω των δικτύων. Δίκτυα που βασίζονται σε ένα ράδιο ηλεκτρικό φάσμα και θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα εκεί υπέρ της καινοτομίας, υπέρ των επενδύσεων για να έχουμε και ανταγωνιστικές αγορές και τελικά ευημερία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ντελκαστήγιο. Βέρα. Η κυρία Σέχνά Λοβά, για ένα λεπτό παρακαλώ. Σα ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ συνάδελφοι. Ομιλώ σαν σκιώδης εισηγήτρια στην Επιτροπή Αναφορών. Οι μεταφορές ε, είναι πρωτοποριακό τομέα στη χρήση των νέων τεχνολογιών μέσω των ευφυών συστημάτων μεταφοράς δεδομένων. Αυτό είναι κάτι το οποίο αυξάνει την ασφάλεια των ταξιδιωτών, καθιστά τις ε, τουριστικές επιχειρηματικές δραστηριότητες πιο αποδοτικές, καλύπτει τις ανάγκες και ε, επίσης ε, θέτει βέβαια το θέμα της προσβασιμότητας των νέων τεχνολογιών, έτσι ώστε να σταματήσουμε να οικοδομούμε νέα εμπόδια. Νομίζω ότι ο εκτός συνδέσεων κόσμος, ο offline world, δεν μπορεί ε, να επιβιώσει μόνος και γι' αυτό χρειάζεται να δικτυωθεί. Ευχαριστώ κύριε Σεγνάλοβα. Για ένα λεπτό τώρα η κυρία Ντίνολφη, παρακαλώ. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Αυτό το θέμα είναι σημαντικό και δεν πρέπει να αφήσουμε την ευκαιρία να χαθεί. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες που προσφέρονται. Και εφόσον πρόκειται για την ψηφιακή εσωτερική αγορά, δεν πρέπει να ξεχνάμε τον πολίτη. Ο πολίτης πρέπει να είναι το επίκεντρο της προσοχής μας. Ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα και ό,τι αναφέρονται στο χάρτη ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αυτά είναι όλα πολύ σημαντικά για την ελευθερία του τύπου, για την ε, ελευθερία ενημέρωσης, κατάργηση διακρίσεων. Πολύ σημαντικά όλα αυτά. Η πραγματική λοιπόν εφαρμογή και υλοποίηση της ψηφιακής εσωτερικής αγοράς μπορεί και να βελτιώσει τη δημοκρατική ζωή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπω όμως δυστυχώς ε, πολύ συχνά να προβάλλονται τα οικονομικής φύσεως θέμα και όχι η ε, δημοκρατική κοινωνική ανάπτυξη. Ευχαριστούμε την κυρία Ντινόλφη. Ακολουθεί για 1,5 λεπτό η συνάδελφος Κόμι. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Επίτροπο. Μετά από αυτή την πολύ καλή δουλειά της ε, κοινοβουλευτικής εργασίας φτάνουμε τώρα στην έγκριση αυτού του ψηφίσματος που είναι ένα πολύ καλό πρώτο αποτέλεσμα. Βεβαίως ποτέ δεν πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι, πρέπει να ζητούμε πάντα κάτι καλύτερο. Πρόκειται λοιπόν για ένα αποτέλεσμα ιδιαίτερο δημοκρατικό. Είναι ο καρπός ε, διαβουλεύσεων, διαπραγματεύσεων και μάλιστα διαπραγματεύσεις ε, όπου εκφράστηκαν πολλά και διαφορετικά συμφέροντα. Ως εισηγήτρια της στρατηγικής ε, για την ενιαία αγορά αγαθών και υπηρεσιών συμμερίζομαι σε μεγάλο βαθμό αυτά που είπε ο κ. Γιούγκε σχετικά δηλαδή με το ότι η ενιαία ψηφιακή κοινή αγορά είναι η προτεραιότητα, μία από τις προτεραιότητες αυτής της Επιτροπής. Και ελπίζω τον δρόμο που έχουμε χαράξει να αποδειχθεί ότι είναι ο σωστός. Πρέπει βέβαια να είμαστε πιο αποφασισμένοι. Έχουμε σημαντικές αλλαγές, ε, το copyright, ε, το ε, διάταξη για το ΦΠΑ, για τα μέσα ενημέρωσης, για τα οπτικοακουστικά μέσα. Δεν θέλω τώρα να σας απαριθμίσω όλα αυτά που αναφέρονται στον κατάλογό μας, αλλά όμως υπάρχουν πολλά θέματα που αναφέρονται στην εμερήσια διάταξη. Εγώ πιστεύω ότι η καθημερινή ζωή, είναι συνδυασμένη με ψηφιακέ εξελίξεις, αυτό αφορά τους επιχειρηματίες και πάρα πολλούς άλλους. Ε, πρέπει λοιπόν να αποδειχθούμε αντάξει του καλέσματος των καιρών. Ε, ο ανταγωνισμός ε, σίγουρα ισχύει και με άλλα κράτη. Εδώ αναφέρομαι κυρίως στις ΗΠΑ που είναι πολύ πιο προχωρημένες. Εγώ λοιπόν θέλω να σας συγχαρώ για τη δουλειά που έχει γίνει και εύχομαι να προχωρήσουμε περισσότερο στο μέλλον. Ευχαριστούμε την κυρία ακόμη. Η συνάδελφος κυρία Στάιλερ έχει το λόγο. Θέλω να πω χρόνια πολλά για τα γενέθλιά της η συνεισηγήτρια την κυρία Γκέπχαρτ που έκανε εξαιρετική δουλειά. Η ενιαία ψηφιακή αγορά έχει ένα τεράστιο δυναμικό. Μιλάμε για εκατομμύρια πολιτών δεκάδες χώρες 450 δις ε, κατέτος κύκλο εργασιών. Πρέπει να είμαστε βέβαιοι βέβαια όταν είναι κανείς στα υψίπεδα της ε, ε, Σκοτίας ή σε άλλες νοτιότερες περιοχές να έχει την δυνατότητα να συνδεθεί. Εδώ πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη και ισότητα στην δυνατότητα πρόσφασης θα πρέπει να μην δημιουργηθεί ένα νεοψηφιακό ρήγμα, θα πρέπει το EICT να είναι διαθέσιμο συνολικότερα. και θα υπάρξουν μέχρι το 2020 και ένα τεράστιος αριθμός θέσεων απασχόλησης που πρέπει να καλυφθεί μια τρίτη ε, βιομηχανική επανάσταση και πρέπει να μην χάσουμε την ευκαιρία. Ευχαριστώ για 1,5 λεπτό, κυρία Νίμπλε, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι. Καταρχά, θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, τι εισηγητρίε, του και όλου και όλου εκείνου που εργάστηκαν για την έκθεση αυτή, που βγήκε πάρα πολύ καλή. Θα ήθελα να συμφωνήσω με την προαλή σα και να ευχηθώ στην κυρία Γκέπχαρτ ε, που έχει γενέθλια χρόνια πολλά. Το 2016 θα πρέπει η ψηφιακή αγορά να κυριαρχήσει, να είναι προτεραιότητα. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε εκείνο το πλαίσιο που θα μας επιτρέψει να αξιοποιήσουμε και να μεταλλευτούμε πλήρω την ευκαιρία στην Ευρώπη. Ξέρετε ότι είναι πολύ μεγάλα τα κοινά που πρέπει να καλύψουμε. 44% των οικοκυριών δεν έχουν γρήγορο ίντερνετ. Άρα καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό και τι κενό πρέπει να καλυφθεί στις υποδομές. Μόνο 14% των μικρομεσαίων κάνουν πωλήσει στο διαδίκτυο ακριβώ διότι υπάρχουν στρεβλώσει και εμπόδια στην αγορά. Θα πρέπει αυτά να έρθουν. Συνάδελφοι αναφέρθηκαν στο γεωγραφικό αποκλεισμό, το geo-blocking. Χρειάζεται και φορολογικό συντονισμό ε, στι καταβολέ ΦΠΑ που πρέπει να απλουστεύονται και να διευκολύνονται και οι πληρωμέ και τα εμβάσματα. Η αντίστοιχη οδηγία, α πούμε, θα πρέπει γρήγορα να εφαρμοστεί για τι πληρωμέ. Κάτι άλλο που έχει σημασία και αυτή είναι η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι θα πρέπει να έχουμε οικοσύστημα για κεφάλαια κινδύνου και για νεοφυείς επιχειρήσεις. Τώρα έχουμε ε, την, ε, ε, της Διεθνής Διάσκεψης που ασχολείται με τις τάσεις και τις εξελίξεις. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Τα νέα μυαλά, τα δημιουργικά μυαλά θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να υλοποιούν τις ιδέες τους στην Ευρώπη και να μην σηκώνονται να φεύγουν στις Ηνωμένες Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Νίμπλερ. Για ένα λεπτό η κυρία Τόγια παρακαλώ. Ehm. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η ανάπτυξη της ψηφιακής αγοράς με τα στάδια τα τόσο σημαντικά τα οποία περιλαμβάνει ο δικός χάρτης θα επιτρέψει να αναπτυχθεί ένας πραγματικά ενιαίος χώρος αγοράς στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Γι' αυτό περιμένοντας το νέο πλαίσιο για τις τηλεπικοινωνίες θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην χάσει την ευκαιρία έτσι ώστε να θέσει σε εφαρμογή τις προτάσεις που κάναμε για τον κανονισμό για τις τηλεπικοινωνίες και να φέρει εις πέρα στις ε, υποχρεώσεις της, ιδιαίτερα σε σχέση με τη χονδρική αγορά. Έτσι μόνο θα μπορέσουμε να σεβαστούμε τις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει στον τομέα του roaming και ταυτόχρονα θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με το geo-blocking, τον γεωγραφικό αποκλεισμό και πώς θα το καταπολεμήσουμε. Στα λίγα δευτερόλεπτα που έχω θέλω να υπογραμμίσω την μεγάλη σημασία που έχει η αγορά αυτή ε, στη συνολικότερη αγορά. Έχουμε πολύ στενές σχέσεις ανάμεσα, διακόπτεται από τον πρόεδρο η κυρία Τόγια. Για 1,5 λεπτό η κυρία Πάουνοβα. Thank you, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έτσι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υπογραμμίσει τον σημαντικό ρόλο που έχει παίξει για την ολοκλήρωση της ψηφιακής αγοράς στην Ευρώπη. Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα είναι αυτό το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Η έκθεση περιλαμβάνει κάποιες χρήσιμες κατευθυντήριες γραμμές, αλλά δυστυχώς δεν είναι πλήρης. θα πρέπει εμείς να ενσωματώσουμε στην online εμπορική δραστηριότητα την εκτός σύνδεσης αντίστοιχη δραστηριότητα έτσι ώστε ε, να θεωρηθεί μια ενιαία αγορά. Αυτό δυστυχώς δεν είναι τμήμα του πρώτου νομοθετικού πακέτου το οποίο έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι η προώθηση των ψηφιακών αγορών στην Ευρώπη θα προωθήσει γενικά και την επιχειρηματικότητα και φυσικά την ολοκλήρωση της ψηφιακής αγοράς και την καινοτομία. Έχουμε διευκρινίσει με τις προτάσεις τις οποίες έχουμε κάνει μέχρι τώρα ότι πρέπει να προωθήσουμε την ψηφιακή αγορά και αυτή έχει μεγάλη σημασία και για την οικονομική ανάπτυξη, για την Ευρώπη την καινοτόμο, την Ευρώπη των νέων, την καλύτερη Ευρώπη και την πιο αποτελεσματική Ευρώπη στην παγκόσμια αγορά. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν τα μέλη της Κοινοβουλευτικής μου Επιτροπής για την προσπάθεια την οποία έκαναν μέχρι τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Για ένα λεπτό η κυρία Κώστα. Η κυρία Κώστα έχει το λόγο. Έχει μεγάλη σημασία να ακολουθήσουμε μια σωστή λογική στον τομέα αυτό, όχι μόνο προς όφελος ε, των ε, καταναλωτών απλά, αλλά του συνόλου των πολιτών θα πρέπει επίσης να εγγυηθούμε για την παρουσία δημιουργικών έργων ε, που ε, εξάπτουν την φαντασία και τη δημιουργικότητα στο διαδίκτυο. Ο ορισμός του αδικαιολόγητου geo-blocking, του γεωγραφικού αποκλεισμού, όπως επίσης και το θέμα ε, του roaming, μια σωστή αντιμετώπιση των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας και των πνευματικών δικαιωμάτων και η σωστή διάκριση ανάμεσα στις ε, ψηφιακές εφαρμογές και υπηρεσίες και τις μη ψηφιακές, ιδιαίτερα στον τομέα της τηλεόρασης, είναι θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στην οδηγία VMS και έτσι θα μπορέσουμε μόνο να προστατεύσουμε την διαφορετικότητα η οποία πρέπει να χαρακτηρίζει την Ευρώπη. Ευχαριστούμε πολύ. Για ένα μισή λεπτό, συνάδελφο κύριο ε, Κόελιο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπο. Ε, νομίζω είναι απόλυτα σαφές ότι η ταχύτατη εξέλιξη έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε και ε, ανταλλάσσουμε εμπορικά προϊόντα στην κοινή αγορά. Αυτή λοιπόν η πραγματικότητα είναι σαφές ότι θα πρέπει να συνοδεύεται και από τη σχετική νομοθεσία για να φέρει όφελος για τις δικές μας τις επιχειρήσεις, για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για τους καταναλωτές πρέπει να προκύψουν ωφέλη. Χαιρετίζω λοιπόν το γεγονός ότι η Κομισιόν όλα αυτά τα έχει αναλάβει ως προτεραιότητα, πολύ καλή στρατηγική της που πρέπει όμως να εξελιχθεί περαιτέρω. Ε, η νομική κατακαιρμάτιση της εσωτερικής αγοράς πρέπει να αποφευθεί, να εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις και μάλιστα εναρμονισμένα. Γιατί αν δεν συμβαίνει αυτό, τότε η Ευρώπη έχει μόνο να χάσει. Πρέπει λοιπόν να κατατεθούν ε, καλές αποτελεσματικές προτάσεις και αυτές ε, σε συνδυασμό με το ψηφιακό περιεχόμενο αλλά και με, τις, ε, και με τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών. Τα δεδομένα, η φορητότητα πέρα από τα σύνορα. Αυτά είναι πολύ σημαντικά. Μια ψηφιακή λοιπόν Ευρώπη που δεν προστατεύει τους πολίτες της είναι μια διχασμένη Ευρώπη. Γι' αυτό η προστασία των δεδομένων είναι πάρα πολύ σημαντική. Πρόεδρος, πολύ ωραία. Πάμε στην επόμενη μιλήτρια που είναι η συνάδελφος κυρία Ουλσκοκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πάρα πολλοί προλαλήσαντες επισήμαναν ήδη ότι η ψηφιακή επανάσταση είναι γεγονός. Ε, οφείλουμε λοιπόν η ψηφιοποίηση αυτή τη στιγμή πρόκειται να αλλάξει τη ζωή μας. Η κοινοποίηση, η δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απευθύνεται στους ε, καταναλωτές ε, Πρέπει να δούμε λιγάκι τις αγορές εργασίας πώς ε, θα πληγούν αυτές. Εκτός αυτού έχουμε και την βιομηχανία ανακύκλωση σε συνδυασμό με την ψηφιοποίηση. Αυτό συνεπάγεται κάποιες ε, προκλήσεις είναι δύσκολο να εφαρμόζονται οι εργασιακές συμβάσεις. Είναι και σαφές το ότι ισχύει crowd working και τηλεεργασία και αυτό συνεπάγεται νέους κινδύνους ε, σωματικούς αλλά και ε, ψυχολογικούς. Οι ευέλικτες μορφές εργασίας μπορούν να είναι ε, θετικές αλλά εμείς δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτή η τάση να οδηγεί σε επισφαλή θέσεις εργασίας. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος ομιλητή για 1,5 λεπτό, ο συνάδελφος κύριος Κέλλη. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ιδιαίτερα για τις νεοπαγείς επιχειρήσεις ε, θα εκμεταλλευτούν την παρουσία της ψηφιακής τεχνολογίας στην ζωή μας. Από τότε που δημιουργήθηκε η Amazon έχουν περάσει 18 χρόνια από τότε που δημιουργήθηκε η Google 12 και εμείς εξακολουθούμε να προσπαθούμε να ορίσουμε σωστά την ψηφιακή αγορά. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι είμαστε πίσω από τις Ηνωμένε Πολιτείες και την Ασία. Το θέμα είναι να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την κατάσταση. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε τα πράγματα. Θα πρέπει να προχωρήσουμε σε εναρμόνιση, να καταπολεμήσουμε τα θέματα του γεωγραφικού αποκλεισμού και να πείσουμε τον καταναλωτή να δείξει εμπιστοσύνη. Εγώ για την Επιτροπή μου ήμουν εισηγητής στα θέματα αυτά και θα πρέπει να εμπνεύσουμε εμπιστοσύνη στους καταναλωτές, να νιώσει ότι ελέγχει την αγορά αυτή και βοηθήσουμε και τις ε, νέες επιχειρήσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Αυτά θα προσθέσουν 450 δις τα επόμενα χρόνια στην ευρωπαϊκή οικονομία. Είναι πολλά τα χρήματα και γι' αυτό πρέπει να εργαστούμε σκλήρα και να ολοκληρώσουμε τον ψηφιακό χάρτη για να γίνουμε πάλι οι πιο αποδοτικοί στον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Για ένα λεπτό ο κύριος Ευχαριστώ. Η ψηφιακή επανάσταση ήδη άλλαξε τη ζωή μας και όπως όλες οι εποχιακού τύπου αλλαγές δημιουργούνται ευκαιρίες και κίνδυνοι. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση αυτή βλέποντας τι δυνατότητες αυξητικές της οικονομικής δραστηριότητας δίνει και διευκόλυνσης προς τους καταναλωτές. Η ψηφιακή τεχνολογία έχει προκαλέσει πάρα πολλές θετικές αλλαγές και στην κοινωνία μας και στην παραγωγική μας δραστηριότητα. Η Ευρώπη πώς ανταποκρίνεται εδώ όταν μιλάμε για τον ψηφιακό κόσμο σκεφτόμαστε το Silicon Valley και όχι την Ευρώπη. Χάρη λοιπόν σε μια σωστή ε, πολιτική, συντονισμένη και ισχυρές επενδύσεις η Ευρώπη θα πρέπει να δείξει τα εξαιρετικά στοιχεία της οικονομικής της δραστηριότητας και να δείξει πόσο σημαντική είναι η ψηφιακή παραγωγή στον τομέα της ποιότητας του πολιτισμού και της φαντασίας. Λοιπόν η Ευρώπη πρέπει να κερδίσει τον χαμένο χρόνο, να ακολουθήσει τον δρόμο της σύγχρονης αντιμετώπισης των προγραμμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα για ένα λεπτό η κυρία Γκάλ Πέλτς παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω καταρχάς ότι θέλω να συγχαρώ τις δύο εισηγήτριες και να ευχηθώ χρόνια πολλά στην κυρία Γκέπχαρτ για τα γενέθλιά της. Είναι καταπληκτική η δουλειά και εξαιρετικά πλήρης η έκθεση και οι δύο εισηγήτριες διακρίθηκαν. Εγώ είμαι σκιώδη συγγήτρια της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Δεν θέλω να επαναλάβω τα όσα υπόθηκαν, να μιλήσω μόνο για τη φορολογία ως προοπτική. Σε αυτό το θέμα έχουμε προχωρήσει πολύ στη ρύθμιση έτσι ώστε να έχουν την απαραίτητη και την αυτονόητη προστασία οι καταναλωτές στην ψηφιακή αγορά. Στο εμπόριο λοιπόν ε, αυτό το ψηφιακό, στην ενιαία ψηφιακή αγορά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και τα φορολογικά σε κάθε ε, ρύθμιση. Να μην έχουμε υπερβολικές ρυθμίσεις, ε, πρέπει να περιοριστεί πολύ η γραφειοκρατία και στηρίζω αυτά που ακούστηκαν η στρατηγική για την ενιαία ψηφιακή αγορά θα πρέπει να ε, συνάδει με την εμπορική πολιτική μας. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό η κυρία Ροζιά. παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τις εισηγήτριες και να συγχαρώ την Εύελιν, όχι μόνο χρόνια πολλά για τα γενέθλιά τη, αλλά ήταν πολύ καλή συνεργασία που είχαμε και πολύ μεγάλη ποιότητα τη συνεργασία μα. Θα ήθελα να μιλήσω εγώ για ένα κλάδο, όλο ιδιαίτερο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι ο πολιτισμό. Είναι γεγονός και το ζούμε όλοι καθημερινά και κάπως μας έχει ενοχλήσει αυτό. Γιατί δεν ικανοποιούμε παντού ε, δωρεάν όλες τις επιθυμίες μας για τον ε, πολιτισμό και σε πραγματικό χρόνο. Θα πρέπει όμως να καθίσουμε να σκεφτούμε πέρα από την ενόχληση τι συνέπειες έχουν οι επιλογές μας. Είναι σωστό δηλαδή να μην έχουμε γεωγραφικό ε, αποκλεισμό, να μην υπάρχει η εδαφικότητα, δηλαδή ένας ε, καλλιτέχνης να μην αμείβεται για τη δημιουργία του, ακόμα και αν αρέσει το έργο του. Σήμερα ε, υπάρχει μια μεγάλη ανισορροπία ανάμεσα στους παρόχους διαχειριστές διαδικτύου και τους ε, δημιουργούς και τους παραγωγούς. Αυτό που διακυβεύεται είναι ο πολιτισμός στην Ευρώπη και αυτή θα πρέπει να είναι η προτεραιότητα όλων μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ραζιέρ. Για ένα λεπτό κυρία Κλούν. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι σκιώδη συγγήτρια της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. Η ψηφιοποίηση, τα εφή μεταφορικά συστήματα είναι το κλειδί για να υπάρχουν αποτελεσματικά συστήματα μεταφορών για τους πελάτες, ε, τους επιβάτες, τις επιχειρήσεις, μικρομεσαίες, ε, νεοφύης, μεγάλες επιχειρήσεις όλους εμάς περιπτώσει που μετακινούν ε, εμπορεύματα και υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Με την ψηφιοποίηση όλα θα είναι πιο αποτελεσματικά και θα καταλήξουν στο να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης. Πολύ σημαντικό αυτό για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις, ε, οι δεσμεύσεις της γραφειοκρατίας κυρίως ε, για τους παρόχους υπηρεσιών. Δεν θα έχουμε τους οδηγούς φορτηγών που θα έχουν να αντιμετωπίσουν όλο αυτό το γραφειοκρατικό φόρτο. Τα αντίγραφα, τα χαρτιά, αυτά κοστίζουν, ε, δημιουργούν αθέμητο ανταγωνισμό και μειώνουν και το δυναμικό για δημιουργία ε, θέσεων απασχόλησης. Άρα δηλαδή πρέπει να καταλήξουμε σε ένα σημείο όπου θα υπάρχουν ρυθμίσεις. Διακόπτη ο Πρόεδρος, ευχαριστούμε κυρία Κλούν. Ε, για ένα λεπτό η κυρία Γιακονσάρη. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω οι συνάδελφοι, οι συγητές ε, εξέτασαν το θέμα εκ του και με μεγάλη περιέργεια θέλω να δω τι θα πει η Κομισιόν για κάποια πράγματα που ακούστηκαν σήμερα εδώ. Πρέπει να συνεχίσουμε την έρευνα, την ανοιχτή έρευνα για να αξιολογήσουμε τις επιπτώσεις της ψηφιακής οικονομίας, στον πολιτισμό, στην οικονομία, στην εκπαίδευση. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και θεωρώ ότι με τον τρόπο αυτό μπορούμε να αποφύγουμε ε, απευκτές επιπτώσεις στην ψηφιακή οικονομία. Χρειαζόμαστε τεχνικές, καλές τεχνικές προδιαγραφές ε, για τον έλεγχο της ψηφιακή αγοράς. Άρα δηλαδή πρέπει να έχουμε κατά νου τα big data, τους αλγόριθμους. Χρειαζόμαστε επίσης ταχύτερες ε, τηλεδιασκέψεις. Πολύ σημαντικό αυτό για την Ευρώπη, για να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτή την τεχνολογική πρόοδο. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Γιακονσάρη, Τώρα λοιπόν για ένα λεπτό η συνάδελφος κυρία Κοράτσα Μπίλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Για να ολοκληρωθεί η ενιαία ψηφιακή αγορά ε, θα πρέπει να έχουμε θάρρος, να ε, ενοχλήσουμε για να δημιουργηθεί αυτός ο μεγάλος αυτοκινητόδρομος, να είναι δωρεάν, παγκόσμιο και ανοιχτό το διαδίκτυο. Υπάρχουν δυνάμεις και χρειάζονται εμπιστοσύνη. Ας ε, ρίξουμε τους φραγμούς, τα εμπόδια και τα σύνορα στην ψηφιακή αγορά. Δεν θα πρέπει ο καταναλωτής να πληρώνει διπλά την ίδια υπηρεσία ανάλογο με το που ζει στην Ευρώπη και η νομοθεσία μας δεν θα πρέπει να είναι ένα άθροισμα 28 εθνικών κανόνων. Χρειάζεται μια ενιαία ψηφιακή ε, αγορά. Υποστηρίζω ε, την έκθεση αυτή απέναντι στους εθνικούς εγωισμούς και προστατευτισμούς. Η Ευρώπη θα πρέπει να έχει κανόνες ε, σύγχρονους ε, και καινοτόμους. Δεν θα προχωρήσει με το να περιχαρακώνεται χρειάζεται διαφάνεια και νέα ψηφιακή αγορά και ελεύθερη ροή των δεδομένων είναι εξίσου σημαντική όπως οι υπόλοιπες τέσσερες ε, ελευθερίες. Ε, θα πρέπει αυτά να συμβαίνουν επιγραμμικά και μη. Και είναι σημαντικό να προχωρήσουμε σε μια συμφωνία για το Safe Harbor και ο χρόνος τελειώνει και δεν θα πρέπει να υπάρξει νομικό κενό. Ευχαριστώ κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Για ένα λεπτό το λόγο έχει ο κύριος ε, Ζωρίνιο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια μεγάλη ενιαία αγορά και θα πρέπει να προσπαθήσουμε για να το πετύχουμε πολύ περισσότερο από ό,τι μέχρι τώρα. Η αγορά αυτή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις βασικές μας αξίες όπως την ελευθερία έκφρασης, την ελευθερία πρόσβασης, την ελεύθερη κυκλοφορία, αγαθών και υπηρεσιών και την προστασία της ασφάλειας των χρηστών. Όλα αυτά είναι τμήμα της ευρωπαϊκής κληρονομιάς και θα πρέπει να μεταφέρουμε εμείς και στην λεγόμενη ψηφιακή ένωση. Η έκθεση κάνει καλές προτάσεις και θα πρέπει να ακολουθήσουμε τις προτάσεις αυτές. Συγχαίρω την εισηγήτρια, θα πρέπει όσο και περισσότεροι Ευρωπαίοι είναι δυνατόν να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και τις ψηφιακές αγορές αυτό θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης, θα βελτιώσει τις γνώσεις και τις ικανότητες των χρηστών και την ψηφιακή <clears throat> καινοτομία. Δεν θα πρέπει να συνεχίσουμε να καθυστερούμε. Θα πρέπει να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατόν. Ευχαριστώ κύριε Τζορίνιο. Και ερχόμαστε τώρα στη διαδικασία Κασιά, αγαπητοί συνάδελφοι. Έχω περίπου 20 συναδέλφους που έχουν ζητήσει το λόγο και μεταξύ αυτών και γραπτές παρεμβάσεις συναδέλφων που ήρθαν στο τέλος της συζήτησης. Θα πρέπει λίγο να τηρήσω το χρόνο. Θα δώσω το λόγο σε συναδέλφους που δεν συμμετείχαν σε άλλες συζητήσεις, σε περιορισμένο αριθμό και μάλιστα συναδέλφους που ήταν παρόντες καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης όσο είχα τη δυνατότητα να το παρακολουθήσω. κυρία Σόιντροβα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Επίτροπε, η ψηφιακή αγορά και το είπαν αυτό πολλοί συνάδελφοι, δίνει τεράστιες ευκαιρίες για την επιχειρηματικότητα στον τομέα και της εμπορίας αγαθών και των υπηρεσιών. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε το κατάλληλο πλαίσιο, έτσι όπως προτείνεται στην έκθεση αυτή, περιλαμβάνονται συγκεκριμένες προτεραιότητες, ε, δύο από αυτές θα τις αναφέρω. Καταρχάς, την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Η πρόσβαση στο περιεχόμενο είναι δικαίωμα των καταναλωτών, οι καταναλωτές όμως έχουν δικαίωμα και στην ποιότητα του περιεχομένου και χωρίς προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Και δεύτερον, η προστασία της παιδικής ηλικίας. Νομίζω ότι είναι χρήσιμο για τα παιδιά το διαδίκτυο, μπορεί όμως να είναι και επικίνδυνος δάσκαλος. Ως εκ τούτου λοιπόν θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες νομοθετικές προτάσεις για την προστασία της παιδικής ηλικίας. Ευχαριστώ κύριε Σόιτροβα. Και τώρα ο κύριος Μπλανκό Λόπεθ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Η ψηφιοποίηση ε, τα έχει κατακλείσει όλα και η Ευρώπη θα πρέπει να αξιοποιήσει όσο γίνεται την ψηφιακή αγορά και να μεταφέρονται περιεχόμενο και ε, να κάνουμε όπως και στο roaming το ίδιο για το γεωγραφικό Ε, Το ραδιοφάσμα ισχύουν τα ίδια. 4.0 είναι πλέον η βιομηχανία, το ίντερνετ των πραγμάτων και δίκτυο ασφαλέ και αξιόπιστο. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τι μικρομέσαίε να αξιοποιήσουν και να εκμεταλλευτούν πλήρω την ψηφιοποίηση. Και θα πρέπει να προστατεύουμε και να προωθούμε τη δική μα πολιτιστική παραγωγή και του δημιουργού. Αλλιώ δεν πρόκειται να συζητάμε για Ευρώπη ξεχωριστή. Μία ευκαιρία έχουμε και η Ευρώπη δεν μπορεί να τη χάσει. Ευχαριστούμε πολύ τον συνάδελφο Πλάνκο Λόπες. Ε, ακολουθεί συνάδελφος Τόμασιτς. Ε, Κύριε Πρόεδρε, η ψηφιακή κοινή αγορά ε, μπορεί να προσφέρει πολλά, να ανάπτυξει το εμπορίο αποτελεσματικότερη διοίκηση. Ενδεικτικά σας ανέφερα κάποια από τα ωφέλη που θα απολαμβάναμε. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να στηριχθεί η καινοτομία και οι επενδύσεις στην τεχνολογία για να επιτύχουμε τους στόχους μας. Εγώ ε, δεν αμφισβητώ τους στόχους, αλλά οι πολιτικοί οφείλουν να κατανοήσουν ότι ε, πρέπει να περιορίσουν τις νομοθετικές ρυθμίσεις για την αγορά και ε, να επιτρέψει να και στην εγκληματικότητα και αυτή πλέον είναι ψηφιακή. Μέσα του διαδικτύου πολλούνται ε, ναρκωτικά, όπλα, προϊόντα μαϊμούδες. Αυτά τα διαδίδουν οι εγκληματικές οργανώσεις. Με την δημιουργία της ψηφιακής κοινή αγοράς θα είναι και πολύ πιο εύκολο να αντιμετωπιστεί η διεθνής εγκληματικότητα. Βεβαίως οφείλουμε να λάβουμε υπόψη μας ότι δεν πρέπει να περιορίζεται η ελευθερία εκείνων ε, που λειτουργούν ομότυπα. Ο συνάδελφος Ρόπε έχει το λόγο. Συνάδελφε Ρόπε, είστε εδώ. Εδώ είμαι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, συνάδελφοι. Τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη στατηγική για την ενιαία ψηφιακή αγορά είναι πάρα πολύ ευπρόσδεκτα. Γίνεται λόγος για δουλειές, για θέσεις εργασίας, για ανάπτυξη εμπορίου, για το φόρο προστιθέμενης αξίας. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία και σημαντικά, αλλά θα ήθελα να σε επιστήσω λίγο την προσοχή στα όσα δεν λέει το κείμενο. Και αυτά είναι οι ανητικές συνέπειες της ψηφιοποίησης των αγορών. Δηλαδή, θα χαθούν, θα εξαφανιστούν τοπικές αγορές, θα μειωθεί η ποιότητα και αν αυτό που μας ενδιαφέρει είναι μόνο ο ΦΠΑ, τότε αυτό θα έχει ανητικές επιπτώσεις σε άλλους κλάδους και τομείς της ανθρώπινης ζωής και δραστηριότητας. Όλα αυτά βέβαια είναι επόμενα και φυσικά ε, ως ε, συνέπειες της παγκοσμιοποίησης. Σωστό είναι αυτό, αλλά αν θέλουμε μια στρατηγική για την ενιαία αγορά, θα πρέπει να κοιτάξουμε να βρούμε έναν τρόπο να θα τον κόσμο για τις επιγραμμικές αγορές, αλλά με το σωστό τρόπο. Με τα λόγου γνώσεως να ξέρει τι αγοράς και τι σημαίνει αυτό για τους λιανοπολιτές και τις μικρές αγορές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ροπέ. Ο κύριος Σόγκορ. Νομίζω ότι ο καθορισμός του τοπίου του ευρωπαϊκού σε σχέση με την ψηφιακή δραστηριότητα είναι κάτι το οποίο είναι ατελές και δείχνει ότι είμαστε μακριά από τις ικανοποιητικές λύσεις και έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις geo-blocking, αποκλεισμού γεωγραφικού και περιορισμών στην φορετότητα των δεδομένων. Σαν αποτέλεσμα οι Ευρωπαίοι καταναλωτές δεν είναι σε θέση να αγοράσουν το περιεχόμενο το οποίο ε, οι γείτονέ του μερικές φορές ε, ε, το κάνουν και πολλές φορές υπάρχουν διαφορές και ανάμεσα σε γειτονικέ όπως είπα χώρες. Είναι λοιπόν πλεονέκτημα για όλους να ανοίξουν οι αγορές έτσι ώστε να γίνει μια πιο πολύγλωση Ευρώπη, μια Ευρώπη με πολλούς πολιτισμούς, της οποίας η επιβίωση, εξαρτάται από την δυνατότητα πρόσβασης και στην ψηφιακή αγορά. Ευχαριστώ κύριε Σόγκουρ. Καπίνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Θέλω να συγχαρώ τους εισηγητές και όσους πήραν μέρος στη σύνταξη της τροπολογίας αυτής. Οι 2.000 τροπολογίες δείχνουν το ενδιαφέρον που έχει προκαλέσει η έκθεση. Η ψηφιακή αγορά είναι ιδιαίτερα σημαντική και νομίζω ότι η εναρμόνιση της νομοθετικής δραστηριότητας είναι προς όφελος των καταναλωτών. Πρέπει να υπάρξουν περισσότερες επίσης δυνατότητες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θυμίζω 100 δις ευρώ δυνητικής ανάπτυξης της οικονομίας για τον τομέα αυτό τον επόμενο, το επόμενο διάστημα. Θα ήθελα λοιπόν να υπάρξει μια ισορροπία ανάμεσα στην χρήση της ψηφιακής αγοράς και την προστασία του καταναλωτή. Δυστυχώς επίσης υπάρχουν προβλήματα προσβασιμότητα στο δίκτυο στις διάφορες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκραπίνη. Ολοκληρώνεται το διαδικασία ΚΑΤΣΔΙ και θα δώσω το λόγο πρώτα στον Επίτροπο κύριο Άνσιπ για να κλείσει η συζήτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για αυτή την επικοδομητική συζήτηση. Ευρώπη μπορέσαμε να οικοδομήσουμε την κοινή αγορά, να καταργήσουμε τα εμπόδια που χώριζαν τα κράτη. Όμως ε, δεν υπάρχει ακόμα η ψηφιακή κοινή αγορά και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η οικονομία μας ε, κάθε μέρα καθίσταται ε, όλο και περισσότερο ψηφιακή. Άρα δηλαδή επανέρχονται τα εμπόδια και αυτά τα προσκόμματα είναι κάθε μέρα ε, όλο και λιγότερο ανυπέρβλητα. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρούμε ότι υπάρχει κάποια πρόοδος. Ήδη τον περασμένο Δεκέμβρη καταθέσαμε δύο προτάσεις. Πρέπει να υπάρχει νομικό περιεχόμενο σε όλες αυτές τις προτάσεις και γι' αυτό καταθέσαμε την πρόταση περί Η δεύτερη πρόταση αφορά τους ε, ψηφιακούς κανόνες για τις ε, συμβάσεις. Ε, τα κράτη-μέλη έχουν 56 διαφορετικές νομοθεσίες για συμβάσεις. Εμείς προτείναμε να υπάρχουν δύο ε, που θα αφορούν στις ε, επιγραμματικές αγορές, επιγραμμικές αγορές ε, με ψηφιακό περιεχόμενο. Η επόμενη πρότασή μας θα κατατεθεί το Φεβρουάριο για τα 700 MHz και ελπίζω και το Μάρτι να μπορούμε να καταθέσουμε την πρώτη μας πρόταση για βιομηχανικούς κλάδους. Θα προτείνουμε ένα βιομηχανικό πακέτο πακέτο το οποίο ε, θα εξετάζει ε, και τις προδιαγραφές της ICT. Τον Απρίλιο θα προτείνουμε ένα άλλο πρόγραμμα δράσης, ε, το Μάιο θα προτείνουμε τη συνεργασία της παραγωγής και των καταναλωτών, το πακέτο ηλεκτρονικού εμπορίου και θα τοποθετηθούμε και για το θέμα του γεωγραφικού αποκλεισμού, geo-blocking. Τον Ιούνιο θα καταθέσουμε δεύτερη πρόταση για το copyright ε, που η πρόταση αυτή τα αφορά την διασυνοριακή πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο αλλά θα ασχοληθούμε και με web libraries, με ε, τα άτομα με αναπηρία. Τον Ιούνιο επίσης ε, θα καταθέσουμε και μία πρόταση για την αναθεώρηση της οδηγίας ε, περί δορυφορικής κάλυψης ε, ε, θα θέσουμε και το θέμα του χρήματος αλλά και τον ρόλο των πλατφορμών το νομικό περιεχόμενο που θα είναι καθοριστικό για το διαδίκτυο Ιούνιο-Ιούλιο θα έχουμε προτάσεις για την κυβερνοασφάλεια αναθεώρηση των κανόνων για τις τηλεπικοινωνίες, ε, για τις υποδομές. Ε, το Νοέμβριο θα τοποθετηθούμε στην ελεύθερη ροή δεδομένων, αναθεώρηση του καθεστώτος ΦΠΑ ε, της ηλεκτρονικής ιδιωτικής σφαίρας και ελπίζω πια το Δεκέμβρη να μην έχουμε νέες προτάσεις για την ψηφιακή αγορά. Προσβλέπω λοιπόν στο να υπάρχει επικοδομητική συνεργασία με εσάς για να ε, επιτύχουμε την ε, ενιαία ψηφιακή αγορά στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πίτροπε. Κύριε Άνση, ακολουθούν τώρα οι εισηγήτριες για να κλείσει συζήτηση. Το λόγο έχει πρώτη κυρία Κάλλας. Δύο λεπτά έκαστε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τη συζήτηση. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το γεγονός ότι συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια τόσε πολλέ κοινοβουλευτικέ επιτροπέ για την εκπόνηση της έκθεσης με γνωμοδοτήσει και τόσοι πολλοί βουλευτέ συμμετείχαν επίσης, ε, εξέφρασαν ανησυχίες και αγωνίες. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένα ζητήματα που ακούστηκαν το πρωί. Πρώτον, θα πρέπει όλοι να κατανοήσουμε ότι το διαδίκτυο δεν είναι ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο. Έχει πάρα πολλά στρώματα και επίπεδα, ε, πολιτιστική πολυμορφία, καινοτομία, έρευνα. Μεταξύ αυτών υπάρχει και το ηλεκτρονικό εμπόριο που έχει τη σημασία του, αλλά δεν είναι το μοναδικό. Ορισμένοι βουλευτέ διαμαρτυρήθηκαν ότι ορισμένα θέματα δεν ε, αντανακλώνται επαρκώ στην έκθεση. Αυτό που έχει σημασία ποιο είναι. Ότι καταφέραμε να βρούμε μια ισορροπία, ότι καλύπτονται όλα τα θέματα και βρήκαμε μια χρυσή τομή στην έκθεση. Ορισμένοι ανησυχούν για την ε, αρχή ε, της μιας φοράς ε, για την προστασία των δεδομένων, once only. Τα δεδομένα, ξέρετε, δεν φυλάσσονται κάπου σε μια τεράστια τράπεζα δεδομένων, αλλά υπάρχουν μικρές τράπεζες δεδομένων οι οποίες μεταξύ τους επικοινωνούν. Αυτό έχει σημασία να το γνωρίζουμε. Και επίση έτσι θα πρέπει να γίνονται τα πράγματα στην ψηφιακή εποχή. Ότι ο κόσμος αναλαμβάνει την ευθύνη των δεδομένων του όταν έρχεται σε επαφή με τις ε, κρατικές αρχές. Και επίση έχει πολύ μεγάλη σημασία ο χρήστη και ο πολίτης να είναι στην καρδιά του συστήματος και να έχει τον έλεγχο των όσων συμβαίνουν. Αυτή η, η οικονομία η συμμετοχική αλλάζει την αγορά και θα πρέπει να δούμε και τα θετικά. Αυξάνει την αυτονομία του κόσμου. Ο κόσμος δεν ε, εργάζεται υπό τον έλεγχο κάποιου, αλλά εργάζεται για τον εαυτό του και αυτό βοηθάει γενικότερα και για την ευημερία και για την πρόοδο. Σας ευχαριστώ όλους και προσβλέπω σε μια καλή συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κάλλας και τώρα η κυρία Κέπχαρτ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και για τα καλά σας λόγια, για τις ευχές για τα γενέθλιά μου. Και νομίζω ότι εδώ βρισκόμαστε εμείς τώρα ε, στην αρχή μιας δουλειάς και όχι στο τέλος. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας για την ενιαία ψηφιακή αγορά και ευχαριστώ πάρα πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας ενημέρωσε για τα επόμενα βήματα και τι μας περιμένει και τι μέλη γενέστε. Όλα αυτά είναι ωραία και καλά. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, ένα θα πρέπει πάντα να έχουμε ξεκάθαρο στο μυαλό μας. Τι θέλουμε, την ε, ενιαία ψηφιακή αγορά μάλιστα. Είναι αυτός σκοπός, όχι. Θέλουμε μια ψηφιακή αγορά ε, στην υπηρεσία των πολιτών, ανδρών και γυναικών. Είτε αυτή είναι παραγωγή, δημιουργή ε, τέχνης, είτε είναι εργαζόμενοι, καταναλωτές, πάροχοι υπηρεσιών. Όλοι αυτοί δραστηριοποιούνται εκεί και θα πρέπει να το έχουμε πάντα στο μυαλό μα και να προσπαθούμε να βγάζουμε πάντα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για να υπάρχει επιτυχία και στον παγκόσμιο ανταγωνισμό να υπάρχει η ευκαιρία να δράξουμε αυτή τη δυνατότητα που διανοίγεται για να υπάρχει μια πραγματική ανάπτυξη με καλές εργασιακές συνθήκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό μας ενδιαφέρει, εκεί θα πρέπει να πάμε και αυτό οφείλουμε να πετύχουμε. Για να τα κάνουμε όλα αυτά θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι και μάλιστα πολύ πιο φιλόδοξοι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το είπαν και ορισμένοι συνάδελφοι προηγουμένω εδώ και από κοινού θα φροντίσουμε να γίνει πραγματικότητα αυτή η προσπάθεια. Τελειώνοντα, θα ήθελα να κάνω και μια παρατήρηση να εξηγούμε για να μην παρεξηγούμε. Η κυρία Τροζίνσκι επέρεται για τις πολλές τροπολογίες που έκανε και στην Επιτροπή και εδώ στην Ολομέλεια. Είναι γεγονός. Αλλά στις συζητήσεις για την έκθεση ήταν απούσα. Δεν την είδαμε σε καμία συνεδρίαση των σκιωδών εισηγητών, ούτε κανένα συνάδελφό της και μην δημιουργούνται τώρα στρεβλές εντυπώσει ότι έχει δουλέψει και πάρα πολύ μάλιστα για ένα θέμα για το οποίο δεν έκανε τίποτα. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ολοκληρώθηκε λοιπόν η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει